Ladies, ladies and gentlemen, I think we should start because it's 10 past. Κυρίες και κύριοι, θα έλεγα να ξεκινήσουμε. Ας επανέλθουμε στη συζήτηση που είχαμε έγιναν συζητήσεις για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε. Σήμερα θα, συζητήσουμε το σχέδιο γράφου γιατί μέχρι στιγμής ασχοληθήκαμε με γενικές δηλώσεις και τώρα θα περάσουμε σε κάτι περισσότερο εξειδικευμένο σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Οι συγητές ασχολούνται με το θέμα της συγκεκριμένη απόφασης θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο που θα πρέπει να καλύψουμε και αρκετά σημεία που θα πρέπει να συζητήσουμε. Δύο λόγια πριν να δώσω το λόγο στους συζητητές. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στις χώρες μας. Διεξήχθησαν εκστρατείες για τη συνθήκη της Λισαβόνας, για την ε, κοινωτική μέθοδο. Και είδαμε ότι ορισμένες χώρες ε, μέλη θέλουν να κινηθεί αυτή η υπηρεσία προς μία κατεύθυνση και αυτό ε, θέτει το θέμα της αξιοπιστίας μας. Θα ακούσουμε λοιπόν την εισήγηση. Νομίζω ότι είχαμε μία πάρα πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά το θέμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και αυτό διαφέρεται και στο έγγραφο που θα συζητήσουμε τώρα. Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τη σύντομη παρουσίαση και τις παρατηρήσεις που κάνατε. Στόχος μας σήμερα είναι να παρουσιάσουμε τα μέλη της ΑΦΚΟ, της Συνταγματικής Επιτροπής, τις προτάσεις τροπολογίας που η ΑΦΕΤ και η ΑΦΚΟ θα πρέπει να προωθήσουν σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου. Όπως γνωρίζετε, οι δύο εισηγητές συνεργαστήκαμε. Οι προτάσεις αυτές για τροπολογία συζητώνται εδώ και ζητηθούν και αργότερα σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Δίχως άλλο, θα είδατε τις τροπολογίες η, τελευταία εκδοχή, η εκδοχή της 3ης Μαΐου του 2010 και ενδεχομένως θα μπορούσα να σας παρουσιάσω αυτές τις τροπολογίες θα το κάνω όμως χωρίς να σας παρουσιάσω τη μία τροπολογία μετά την άλλη, γιατί γι' αυτό θα πετηθούν αρκετές ώρες. Θα τις συγκεντρώσω λοιπόν, τις ε, τροπολογίες, κάτω από συγκεκριμένους τίτλους. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες. Το πρώτο μέρος των τροπολογίων αφορούν θεσμικές ε, πτυχές του σχεδίου απόφαση. Όπως γνωρίζετε, θέλαμε η Ευρωπαϊκή αυτή υπηρεσία εξωτερικής δράσης να είναι συνδεδεμένη με την Επιτροπή από την άποψη τη διοικητική και από την άποψη του προπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα πρέπει να αποτελέσει μέρο του τμήματο 3 του Γενικού Προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στι τροπολογίε, στο εκτιμώντα 1 και στο εκτιμώντα 7, και η τροπολογία στο άρθρο 1-2 είναι οι τροπολογίες που έχουμε προσθέσει για να λάβουμε υπόψη μας το σημείο αυτό, για να εξετάσουμε τη θεσμική πτυχή της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, αλλά και για να την προσαρτήσουμε, να τη συνδέσουμε με την Επιτροπή σε επίπεδο οργανωτικό, διοικητικό, αλλά και από άποψη προπολογισμού. Το δεύτερο μέρος των τροπολογιών αφορούν το κατά πόσον είναι υπόλογη υπηρεσία στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρότασή μας είναι ο ύπατος εκπρόσωπος και ο αντιπρόεδρος και της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να είναι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ό,τι αφορά πολιτικά θέματα αλλά και σε ό,τι αφορά θέματα προϋπολογισμού. Θα το δείτε αυτό στις τροπολογίες, το εκτιμώντας 5 και στο άρθρο 1.3α. Είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά το θέμα της πολιτικής ευθύνης θα πρέπει να το να καταστήσουμε σαφές το τι εννοούμε με το ότι η πολιτική υπευθυνότητα και αυτό θα είναι σε ένα μνημόνιο που θα πρέπει να συμπεριλάβουμε σε αυτή την απόφαση. Το τρίτο μέρος των τροπολογιών αφορούν την πολιτική εκπροσώπηση την, ε, της ΥΠΑ ΕΕ, της εκπροσώπου και την Προέδρου. Όπως γνωρίζετε, Είμαστε υπέρ του να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο ορισμένοι επίτροποι έτσι ώστε η ύπατη εκπρόσωπος να μπορεί να εκπροσωπείται από μια σειρά από εκπροσώπους, ε, Επίτροπο για Ανάπτυξη, Συνεργασία, Πολιτική Διετίασης, ε, ε, Βοήθειας κτλ, Σχετικής Βοήθειας κτλ. Όλα αυτά τα συμπεριλάβαμε στο σχέδιο απόφασης και προβλέπουμε επίσης μία σειρά από ε, αναπληρωτές. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στην τροπολογία μας το άρθρο 2α του σχεδίου απόφασης. Το τέταρτο μέρος των τροπολογιών αφορά το συντονισμό της πολιτικής στο εσωτερικό της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Αν έχετε την εκπρόσωπο, αν έχετε ένα αριθμό ε, ε, επιτρόπων που μπορούν να εκπροσωπήσουν τον ύπατο εκπρόσωπο για θέματα κοινοτική αρμοδιότητα και παράλληλα υπάρχουν και ορισμένοι αναπληρωτέ που μπορούν να την εκπροσωπήσουν. Επίση, αλλά και παράλληλα στην ε, κοινή πολιτική ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, είναι αναγκαίο αυτό να συνδυαστεί στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Αρχικά θεωρήσαμε ότι ήταν καλή ιδέα να εντάξουμε ένα φορέα συντονισμού πολιτικής. Αυτό όμως είναι μια καινούρια οργάνωση δημιουργούμε μια καινούργια οργάνωση μέσα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία και τελικά η πρότασή μας είναι να προβλέψουμε ένα μηχανισμό συντονισμού της πολιτικής στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η διασύνδεση ότι υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ της υπηρεσίας κοινωνικής δράσης και της Επιτροπής και αυτή η σχέση ενδυναμώνεται και υπάρχει και μια συνοχή μέσα σε αυτή την υπηρεσία. Δηλαδή, οι ύπατη εκπρόσωπο μαζί με τους αναπληρωτές και τους ε, ε, επιτρόπους κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Γι' αυτό προβλέπεται ένας μηχανισμός συντονισμού της πολιτικής. Δεν, θα δημιουργηθεί <clears throat> μια καινούρια οργάνωση. Ένας μηχανισμός στα πλαίσια της υπηρεσίας και αυτό αναφέρεται στην τροπολογία στο άρθρο 2β. Η πέμπτη πρόταση στην ε, τροπολογίες μας είναι, όπως γνωρίζετε, αφορά την αντικατάσταση στο σχέδιο απόφαση στο Γενικό Γραμματέα με ένα γενικό διευθυντή που διορίζεται από το, την ύπατη εκπρόσωπο. Γιατί θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης ε, είναι μια υπηρεσία, δεν είναι ένας θεσμός και συνεπώς θα πρέπει να οργανωθεί η διαχείριση στο εσωτερικό αυτής της υπηρεσίας με έναν γενικό διευθυντή. Και αυτό προβλέπεται στην τροπολογία στο άρθρο 4.1. Οι επόμενες τροπολογίες αφορούν τον συντονισμό μεταξύ της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της άλλες εξωτερικές πολιτικές της Επιτροπής. Δηλαδή, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αποτελείται πρωτίστως από τους επιτρόπους, την είπατε εκπρόσωπο και τους αναπληρωτές, αλλά υπάρχουν και άλλες εξωτερικές πολιτικές στην Επιτροπή. υπάρχει το ε, θέμα των ε, κλιματικών αλλαγών. Συνεπώς προβλέπεται στην υπηρεσία αυτή ένα interface, μια ενδιάμεση υπηρεσία η οποία συνδέει τις ε, υπηρεσία αυτή με τις, άλλε με τις άλλες αυτές υπηρεσίες που βρίσκονται κυρίως μέσα στην Επιτροπή και που ασχολούν άλλα θέματα που αφορούν εξωτερική δράση. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι αναγκαίο όλα αυτά τα θέματα να ενταχθούν στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν ενδιάμεσο φορέα έτσι ώστε να υπάρχει συνοχή μεταξύ των απόψεων που υιοθετούνται μεταξύ του ενός τμήματος και των άλλων. Των απόψεων δηλαδή που υιοθετούνται από την υπηρεσία εξωτερική δράσης. Η δημιουργία λοιπόν αυτού του ενδιάμεσου φορέα προβλέπεται από την τροπολογία για το, στο άρθρο 4 σημείο 2. Επόμενο σημείο στις τροπολογίες αφορά την αντιμετώπιση, τη διαχείριση της κρίσης, των κρίσεων στο μέλλον. Αυτό που προτείνουμε είναι να συμπεριληφθούν όλες οι σχετικές υπηρεσίες που ασχολούνται με το θέμα της διαχείρισης κρίσεων σε μία και μοναδική διεύθυνση. Μία και μοναδική διεύθυνση, λοιπόν, η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Δεν θα είναι κάτι εκτός της υπηρεσίας και της δράση, δεν είναι κάτι που θα εξαρτάται από την υπατή, από την υπατή εκπρόσωπο, ή θα είναι μια διεύθυνση στο εσωτερικό στα πλαίσια της υπηρεσία και ζωητικής δράσης. Είναι βεβαίως σαφές ότι όταν έχουμε με επιχειρηματικές αποστολές η ύπατη εκπρόσωπος θα έχει, θα παίρνει την τελική απόφαση σε ό,τι αφορά τις σχετικές υπηρεσίες. Και αυτό προβλέπεται στην τροπολογία μας στο άρθρο 4.3. Συνεπώς, το όλο θέμα για τη διαχείριση των κρίσεων έχει μεταγραφεί σε ένα, μια τροπολογία στο 4.3. Το επόμενο θέμα είναι το θέμα των αντιπροσωπιών θα δίνονται εντολέ, θα δίνονται οδηγίε από την ύπατη εκπρόσωπο και προβλέπουμε ότι σε περίπτωση σύγκρουσης θα διεξάγεται μία συζήτηση μεταξύ της ύπατης εκπροσώπους ε, και όλες οι διαφωνίες θα επιλύονται στο εσωτερικό της Επιτροπής από το Κολέγιο των Επιτρόπων. Αυτός ο μηχανισμός έχει μεταφερθεί, έχει μεταγραφεί σε μία τροπολογία στο άρθρο 5.3. Επόμενο θέμα αφορά το προσωπικό. Όπως γνωρίζετε, το προσωπικό για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι κυρίω άτομα υπάλληλοι τη Επιτροπή και του Συμβουλίου και ορισμένοι προσωρινοί υπάλληλοι που προέρχονται από τις χώρες μέλη. Στο σχέδιο απόφασης υπάρχει και η ιδέα του να χρησιμοποιηθούν εθνικοί εμπειρογνώμονες. Λέμε ότι αυτό θα πρέπει να περιοριστεί στο στρατιωτικό προσωπικό που απαιτείται για, την διαχείριση, για τις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. Αυτό και πάλι έχει μεταφερθεί σε μια τροπολογία στο άρθρο 6, 6.1β. Επόμενο θέμα, η εξισορρόπηση σε ό,τι αφορά την ε, ε, γεωγραφική της χώρες και τα, ε, το, το, τα φύλλα. Ε, προσώπηση, προσώπηση ανδρών και γυναικών άρθρο 6.6. Επόμενο θέμα, όπως γνωρίζετε, αφορά την αναλογία πόσοι προέρχονται από τις χώρες μέλη, πόσοι προέρχονται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, ένα τρίτο από τις χώρες μέλη, αλλά πάνω από το 90% από την Επιτροπή. Αυτό είναι ο στόχος του Κοινοβουλίου και αυτό οδήγησε στη σύνταξη μιας τροπολογίας το άρθρο 6.10. Ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός είναι το επόμενο θέμα στις τροπολογίες. Κατά την άποψή μας, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης έχει μόνο ένα διοικητικό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνεται στο κεφάλαιο 5 του προϋπολογισμού. Ξέρετε, τα διάφορα κεφάλαια του προϋπολογισμού το κεφάλαιο 5 αφορά τα δίκη, τις διοικητικές δαπάνες και αποτελεί και μέρος του τμήματος 3. Ε, κεφάλαιο 5 ε, σημείο 3. Είναι το σημείο που εντάσσεται ο προπολογισμό υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Αυτό αναφέρεται στο εκτιμώντας 7 και στο άρθρο 7. Στο 1. Σε δύο σημεία αναφέρεται. Περνάμε το σημαντικό θέμα του προγραμματισμού του προγραμματισμού της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Πώς θα επιληφθούμε αυτού του θέματος. Όπως γνωρίζετε, η θέση του Κοινοβουλίου είναι να υπάρξει ένας σαφής καθορισμός του ρόλου στον προγραμματισμό και αυτό σε σχέση με τις άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, να δούμε ποιος είναι υπεύθυνο για τις λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από τις εξωτερικές δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, κατ' ουσία αυτό που προβλέπουμε στις τροπολογίες μας είναι ότι η, εξωτερική, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα εμπλακεί στις φάσεις 1 έως 3 του προγραμματισμού και στις επόμενες φάσεις εφαρμογής του προγραμματισμού ή αρμοδιότητα των άλλων υπηρεσιών της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια ότι στην πρότασή μας και αυτό είναι μια αλλαγή από το σχέδιο απόφασης, δεν υπάρχει διαχωρισμός, για παράδειγμα, με, ε, στην ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ οριζόντια θεματικά θέματα και γεωγραφικά θέματα και καθήκοντα. Όλα αυτά λοιπόν παραμένουν σε έναν κύκλο του προγραμματισμού. Γιατί στην πρόταση, όπως την έχουμε μπροστά μας σήμερα, στην πρόταση του Συμβουλίου, τα οριζόντια θεματικά θέματα αφορούν την Επιτροπή, μετά περνάμε στα γεωγραφικά θέματα και μετά για θέματα εφαρμογής και πάλι αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες ε, της Επιτροπής. Και κατά την άποψή μας και δίχως άλλο κατά την άποψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, γιατί ο κύριος Ζαμπρόκο και εγώ ε, πήγαμε στην Επιτροπή για να ακούσουμε την άποψή τους σχετικά με αυτό το θέμα, τη στάση τους σε ό,τι αφορά την πρόταση και καταλήξαμε ότι υπάρχει μια γενική εντύπωση ότι θα πρέπει να αποφύγουμε αυτό τον, ε, τη διαφοροποίηση μεταξύ οριζόντιων και διαγραφικών θεμάτων ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Αυτό που προβλέπουμε είναι ότι όλες οι φάσεις από ένα ε, ως τρία συγκεντρώνονται στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και μετά η εφαρμογή, την εφαρμογή την αναλαμβάνουν οι άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής. Και οι δύο αυτές αρχές περιέχονται στις τροπολογίες στο άρθρο 8.1 και στο άρθρο στο 8.2, στις του 8.2. Αυτό που προβλέπουμε επίσης είναι το προνόμιο των αρμόδιων επιτρόπων, προνόμιο που θα συνεχίσει να υφίσταται, δηλαδή δεν χάνουν καμία από τις αρμοδιότητες τους σαν αποτέλεσμα της δημιουργίας της υπηρεσίας και δράσης και αυτή η αρχή έχει συμπεριληφθεί τη μεταγραφή σε μία τροπολογία στο άρθρο 8.2. Τέλος. Έχουμε το θέμα της πρόσβασης στα έγγραφα. Όπως γνωρίζετε, η πρόσβαση σε τα έγγραφα ε, θα πρέπει επίσης να προβλέπετε αυτό σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο και έχει προβλεφθεί μία τροπολογία στο άρθρο Κύριε Πρόεδρε, έκανα μία σύντομη ανασκόπηση του όλου πακέτου των τροπολογιών. Δεν σας περιέγραψα λεπτομερώς την κάθε τροπολογία. Ε, τα εξέτασα ένα θέμα, κεφάλαιο. Κατά την άποψή μου, καταφέραμε να μεταφέρουμε το αρχικό non-paper και μετά το έγγραφο που σας υποβάλαμε ο κύριος Μπρόκ και εγώ, που υποβάλαμε στην Επιτροπή σας, βεβαίως είναι σαφές ότι αν το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι δύσκολο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και να δεχτεί τις τροπολογίες μας, δίχως άλλο. Ε, ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμο να προβλέψουμε άλλε τροπολογίε. Αυτό βεβαίω εξαρτάται από το Συμβούλιο, αν θα μπορέσει να συμφωνήσει ή όχι. Λέγοντα νέε τροπολογίε, εννοώ ότι θα πρέπει τα πάντα να επανέλθουν στην Επιτροπή. Αυτό είναι μια εναλλακτική λύση, αν θα ακολουθήσουμε τη γραμμή του Συμβουλίου. Αν θέλουμε μια φιλόδοξη υπηρεσία εξωτερική δράση που θέλουμε να έχει τόσους δημόσιους ε, υπαλλήλου που θα ασχολούνται με την πολιτική γυπνία με τη συνεργασία, με την ανάπτυξη κτλ. Αλλά βεβαίως αν υπάρχουν προβλήματα για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, τότε, δηλαδή η σύνδεση της υπηρεσίας με την Επιτροπή δεν το αποκλείω να χρειαστεί να σκεφτούμε τις τροπολογίες αυτές σε, αυτό το, σε αυτή την Επιτροπή και να κινηθούμε προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Ναι, ενδεχομένω θα πρέπει να μεταφέρουμε όλες αυτές τι αρμοδιότητε προ την Επιτροπή. Αυτό όμω είναι κάτι που αφορά το μέλλον. Αυτή είναι μία παρατήρηση που απλώς ήθελα να κάνω στο τέλος της παρουσίαση αυτών των τροπολογιών, κύριε Πρόεδρε. Είναι λοιπόν το λόγο στον εισηγητή, τον ε, κύριο Έλμα Μπροκ. Κύριε Πρόεδρε, ε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα το σημαντικό σε αυτά που είπε ο προλαλής σας, συνάδελφος, και θέλω απλά να επισημάνω ότι πέρα από το έγγραφο επί το καλούμε θα να αποφανθούμε και βεβαίως ε, θα υπάρχουν και σχετικές ε, ψηφοφορίες για τους κανονισμούς περί προσωπικού και περί προεπολογισμού. Σίγουρα θα γίνουν αυτές οι ψηφοφορίες, αλλά αυτές ε, δεν θα ενταχθούν στον κανονισμό και αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό γιατί θα πρέπει πρώτα απ' όλα να καθορίσουμε προδιαγραφές όσον αφορά το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαπραγματευόμαστε με την Κομισιόν. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχει και μία συμφωνία που θα παρουσιαστεί στην κυρία Άστον μια συμφωνία που θα αφορά στα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβουλεύσεων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει στα κράτη-μέλη. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε μια καινούργια αρχή και από την αρχή πρέπει να θέσουμε κάποιους ε, κανόνες. Ε, θα ήθελα απλά να σα αναφέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Παραδείγματο χάρη, ω ε, Κοινοβούλιο, έχουμε κάποια δικαιώματα για να ρυθμίσουμε τα οικονομικά των αντιπροσωπιών. Έχουμε επίση κάποια δικαιώματα για τη σύναψη συμβάσεων και συμφωνιών. Και τίθεται το εξή ερώτημα. Όσον αφορά στις εντολές που δίδονται για αντιπροσωπείες, για επισκέψεις, το Κοινοβούλιο θα εισακούεται, θα εκφράζει την άποψή του. Αυτό λοιπόν το θέμα πρέπει να ρυθμιστεί γενικότερα, οριζόντια. Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμιστεί ε, ποιοι άνθρωποι μπορούν να αναλαμβάνουν τέτοιου είδου αποστολέ. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πρακτική φύσεως θέματα, όπως ε, παραδείγματο χάρη και το θέμα του στρατού, των επεμβάσεων. Οι πρέσβεις, οι ειδικοί εκπρόσωποι, αυτοί πρέπει να παρουσιάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει κάπως να διασφαλιστεί ότι αυτή η υπηρεσία είναι και μια υπηρεσία που εκπροσωπεί το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εκ τούτου όλους τους φορείς. Άρα δηλαδή θα πρέπει να παρουσιάζεται στο Κοινοβούλιο. Και θέλω να σας αναφέρω και εδώ κάποια παραδείγματα. Υπάρχει και άλλο ένα επίπεδο διαπραγματεύσεων, όπου αυτό ισχύει εν μέρη και για τα δημοσιονομικά, τα δημοσιονομικά αναφέρεται ότι αυτά τα θέματα, τα δημοσιονομικά, πρέπει να ρυθμίζονται μέσα στον ε, σχετικό κανονισμό. Αλλά ε, σας επαναλαμβάνω, και εκεί πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα της εκπροσώπησης. Αυτό το έγγραφο της ε, κυρίας ε, Άστον, το έγγραφο του Συμβουλίου δεν αρκεί αν δεν έχουν πληρωθεί και αυτές οι προϋποθέσεις που σας ανέφερα. Και εδώ λοιπόν πρέπει να ρυθμιστούν κάποιες ε, προϋποθέσεις έτσι ώστε στα γενικής φύσεως θέματα να βρούμε κάποια λύση. Και αυτό έχει σχέση με το συντονισμό της ε, πολιτικής ε, εκπροσώπησης. Τούτο πάλι έχει σχέση με τα δημοσιονομικά δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την πολιτική ευθύνη ποιος την αναλαμβάνει σε περίπτωση που απουσιάζει η κυρία Άστον. Και αυτό το θέμα τίθεται στις διαπραγματεύσεις. Θα λοιπόν για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω ότι οφείλουμε να έχουμε κάποιες επίσημες διαπραγματεύσεις ε, όταν θα κατατεθεί η έκθεση του κυρίου Φερχόφστατ και η δική μου, η κοινή μας έκθεση. Θα τεθούν λοιπόν όλα τα θέματα επιτάπητος και το θέμα του κανονισμού προσωπικού. Ως εκ τούτου θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα αναφέρεται στο δικό μας το έγγραφο για την απόφαση του Συμβουλίου αφενός και αφετέρου τι θα πρέπει να προσθεθεί στον ε, δημοσιονομικό κανονισμό και στον κανονισμό περί προσωπικού. Ή, αν θέλετε, τι πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά και δύο σε αυτά τα τελευταία δύο θέματα. Ε, εδώ θα έχουμε διαβουλεύσει με τον κύριο Ραπ και με τον κύριο Νοτέρη για να δούμε ποιο θα είναι από τακτική πλευρά ο καλύτερο δρόμος. Ο κανονισμός του Συμβουλίου, στη τελική ανάλυση, μπορεί να τροποποιηθεί εκ νέου από το Συμβούλιο. Ο δημοσιονομικός κανονισμός ε, και ο κανονισμός περί προσωπικού μπορούν να τροποποιηθούν μόνο μέσα από τη διαδικασία της συναπόφασης, όχι με απλή απόφαση του Συμβουλίου. Άρα δηλαδή εμάς μας συμφέρει στα τελευταία δύο να θεσπίσουμε κάποια θέματα για να μην μπορούν να ε, τροποποιηθούν χωρίς τη δική μας την τοποθέτηση. Νομίζω λοιπόν ότι θα βρούμε κάποια λύση οι δύο εισηγητές και οι δύο επιτροπές και θα μπορέσουμε τελικά να καταθέσουμε μια πρόταση η οποία πρόταση ε, θα θεωρείται ότι εκφράζει συνολικά τη δική μας θέση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Σεβερίν. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι οι προσπάθειε των δύο συγητών το να συνδυάσουν ε, τα δύο θέματα και να βρεθεί μια κοινή άποψη, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σωστό. Εγώ πιστεύω αυτά που ελέγχθησαν από τον κύριο Μπροκ ε, εκπέμπουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Δηλαδή, όλοι οι συγητές από τις διάφορες επιτροπές θα πρέπει να καταλήξουν σε μια κοινή θέση. Και αυτό το μήνυμα οφείλουμε να το διαβιβάσουμε στο Συμβούλιο, ότι δηλαδή είμαστε όλοι ενωμένοι στο να ε, εκπροσωπούμε μια κοινή θέση. Και βεβαίως θα πρέπει η θέση αυτή να βασίζεται στις προτάσεις που μόλις τώρα ακούσαμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν τέσσερις ε, λέξεις κλειδί, ε, λέξεις σημαντικές, πρέπει να τις ελέγξουμε όσον αφορά τις προσπαθίες μας. Διαφάνεια, απόδοση λόγου σε θέματα δημοσιονομικά και άλλα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι οτιδήποτε υπάρχει στα έγγραφά μας και οτιδήποτε υπάρχει στις αξιολογήσεις του Συμβουλίου και της Κομισιόν, οτιδήποτε λοιπόν θα πρέπει να ελέγχεται κάτω από το πρίσμα αυτών των τεσσάρων λέξεων κλειδί. Δηλαδή, είναι διαφανείς οι θέσεις, επιτρέπουν να υπάρχει απόδοση λόγω, όπως είπα, με σωστό τρόπο και από δημοσιονομικό ε, πρίσμα και από άλλο. Αυτές οι προτάσεις προσφέρουν ε, την ελπίδα για συνένεση, για συνοχή, αποτελούν μια καλή βάση για αποτελεσματικότητα. Αν λοιπόν η απάντηση σε αυτά τα θέματα είναι καταφατική, τότε νομίζω ότι πράγματι καταλήξαμε σε μια ικανοποιητική λύση. Αλλιώ θα πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα. Και τώρα επιτρέψτε μου κάποιε ε, πολύ συγκεκριμένε παρατηρήσει που αφορούν ε, στην έκθεση του κ. Φερχόφστατ. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι αυτή η φόρμουλα που προσαρτάται στην Κομισιόν νομίζω ότι είναι ικανοποιητική. Δηλαδή, είναι ικανοποιητική γιατί πράγματι χρησιμοποιείται στι ε, διεθνεί σχέσει σε διάφορου τομεί. Ως εκ τούτου, για πάρα πολλούς ε, αυτή η διατύπωση είναι ικανοποιητική, ε, λέει κάτι, υπάρχει σχετική νομολογία, υπάρχει μια πρακτική, άρα να ε, διατηρήσουμε αυτή τη διατύπωση. Και αυτή η διατύπωση υπογραμμίζει τον ιδιότυπο χαρακτήρα της υπηρεσία εξωτερικής δράση και βοηθά και εμά να κατανοήσουμε τι ακριβώ σημαίνει αυτό το sui το ιδιόμορφο αν θέλετε. Αυτό το ιδιόμορφο θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Οφείλουμε λοιπόν να το ορίσουμε επακριβώς, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι πράγματι αφορά αυτό που επιθυμούμε και όχι κάτι άλλο. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τον ε, μηχανισμό συντονισμού πολιτική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι εδώ Έχουμε δύο δυσδιάστατους μηχανισμούς συντονισμού. Ο ένας είναι εσωτερικός, όπως ελέγχθη, και ο δεύτερος αφορά το συντονισμό ανάμεσα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ε, θα ήθελα μετά να δώσω το λόγο στον κ. Φεχόφτατ. Εγώ το μόνο που θέλω να προτείνω εδώ αφορά στο 2β νέο. Εκεί λοιπόν να πούμε στην τελευταία πρόταση ότι οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο και άλλοι επίτροποι θα μπορούν να αποτελούν τμήμα αυτού του μηχανισμού. Ε, θα ήταν πολύ πιο ευέλικτο αν πούμε όχι άλλοι επίτροποι, αλλά άλλοι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών. Γιατί νομίζω ότι είναι σωστό σε αυτό το μηχανισμό συντονισμού να έχουμε ως το δυνατόν περισσότερους μπορούν να συμβάλλουν και που μπορούν να λάβουν και αποφάσεις ε, ε, μάλλον που μπορούν να υιοθετήσουν αυτό τον ε, μηχανισμό συντονισμού. Εδώ πρόκειται για θέμα περισσότερο ευελιξία και όχι ουσία. Ε, διαχείριση κρίσεων από την Επιτροπή και μέσα στην Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, πολύ σημαντικό αυτό και σωστό. Και τέλο, δεν θέλω να σχολιάσω όλα τα υπόλοιπα. Επί της ουσίας συμφωνώ. Ίσως κάποιες μικρές αλλαγές να προταθούν. Πάντως, κατά τη δική μου άποψη, και νομίζω ότι ο συνάδελφος ο κύριος Γκουαλτιέρη θα προσθέσει κάτι σημαντικό επ' αυτού όσον αφορά στον προπολογισμό. Αλλά για μένα ο προπολογισμό είναι θέμα κλειδί. Και εγώ, ενώ στα άλλα θέματα θεωρώ ότι προχωρήσαμε ικανοποιητικά, εδώ δεν νομίζω ότι προοδέψαμε, ότι προχωρήσαμε. Ίσως κάπως, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Διότι ο προπολογισμό αποτελεί την σύνθεση των πολιτικών αποτελεί την συνθετική έκφραση των προγραμμάτων και των πολιτικών και παράλληλα αποτελεί ένα εχέγγυο ότι ε, τα προγράμματα πράγματι θα υλοποιηθούν. Ως εκ τούτου χαιρετίζω αυτήν την ιδέα της ε, θεματικής, γεωγραφικής, λειτουργικής ε, συνοχής, αλλά πρέπει να υπάρχει αυτό που με τον κύριο Ρομπέρτο Κουαλτιέρη θα αποκαλούσαμε σταθεροποιημένο ή ενοποιημένο προπολογισμό. Ενοποιημένο προπολογισμό. Νομίζω ότι ορισμένα θέματα ε, θα πρέπει ε, να τα αναλάβουν άλλοι φορεί στο πλαίσιο της πολιτικής τους, αλλά δεν υπάρχει ούτε διαφάνεια, ούτε απόδοση λόγου, εάν ο προπολογισμό απλά κατακαιρματιστεί και δεν μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα του προπολογισμού, όχι μόνο για τα διοικητικά, αλλά για τα πολιτικά και λειτουργική φύσεως θέματα. Ε, έτσι λοιπόν, για να είναι άνθρωποι υπόλογοι, για να μπορούμε να έχουμε έτσι μια πολιτική εποπτεία, για να μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πράγματι η συνοχή, η θεωρητική μεταφράζεται σε πρακτική συνοχή των φορέων, χρειαζόμαστε έναν ενοποιημένο προπολογισμό οργανισμό ο οποίος ε, θα συγκεντρώνει τα πάντα. Και όχι να υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ξέρετε όμως αυτές οι δραστηριότητες ε, είναι εκτός των κοινοτικών εκείνων πράξεων ε, τις οποίες ελέγχει το Κοινοβούλιο. Όχι, θα πρέπει να μπορούμε μόνοι μας να κατανοήσουμε πώς ακριβώς τούτο συμβαδίζει με το σύνολο του προϋπολογισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι οι συγητές πρέπει να βρουν κάποια λύση για να είμαστε και εμείς σίγουροι ότι τελικά μπροστά μας ως βουλευτές θα έχουμε έναν ενοποιημένο προϋπολογισμό, έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα μιλάει για το σύνολο των εξωτερικών δράσεων που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι λοιπόν θα μπορούμε να εγκρίνουμε και εμείς αυτόν τον προϋπολογισμό και να παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται ο προϋπολογισμός. Γιατί αν δεν γίνει αυτό φοβάμαι ότι θα έχουμε μία μερική άποψη για την οικονομική υποστήριξη των πολιτικών που επιθυμούμε να προάγουμε. Και επίσης, λόγω αυτού δεν θα μπορούμε να αξιολογήσουμε το κατά πόσο μια πράξη είναι συνεπής ή όχι με την υπόλοιπη πολιτική μας. Και βεβαίως δεν θα μπορέσουμε να ζητήσουμε την απόδοση λόγου από εκείνους οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση του προπολισμού και την εφαρμογή των πολιτικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, νομίζω έχουμε πάει καλά. Η πρόοδος συνίστερα ακριβώς στις αλλαγέ που έχουμε επιφέρει. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο στόχο μας και αυτό είναι καλό. Και επιπλέον, όλα αυτά αποτελούν μια αποτελεσματική διαδικασία συναπόφασης. Δηλαδή η απόφαση αυτή μαζί με τους δημοσιονομικούς κανόνες, μαζί και με το MOU, το Μνημονίο Συνεργασίας, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά μαζί. Από εδώ και πέρα πρέπει να βοηθήσουμε την Κάθριν Άστον να συντάξει αυτό το μνημόνιο κατανήσεων, μνημόνιο συνεργασία μεταξύ της Ιδίας και ημών με ΙΤΑ. Σε αυτή τη διαδικασία εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό εάν το χρειαστούν και οι συγητές βεβαίως. Θεωρώ ότι τόσο ποσοτικός όσο και ποιοτικός ακούστηκαν αξιολογότερες θέσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση. Με σεβασμό και την ισορροπία εξουσιών και αρμοδιορίτων. Τώρα, όσον αφορά το ίδιο το κείμενο, Δεν ξέρω αν έχει τόση σημασία και έννοια να απαιτήσουμε ε, καθηνάστον να είναι σε κάθε περίπτωση στο Κοινούλιο. Το Συμβούλιο νομίζω ότι θα αντιδράσει γιατί καθηνάστον σε αυτό αναφέρεται. Μπορούμε παρόλα αυτά να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία και ως προς αυτό το ερώτημά μου είναι θα υπάρχει πρόβλημα και ποιο είναι αυτό. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία πλέον. Και ποια είναι επιτέλους τα σημεία στα οποία διαφωνούμε τι μας εμποδίζει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ίσως οι συζητές θα μπορούσαν να απαντήσουν το με αυτό και να μας πούν σε ποιο σημείο βρίσκονται ακριβώ οι διαπραγματεύσει τους με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Τέλος, όπως έχω δηλώσει κατά επανάληψη και πριν τις Βρετανικές εκλογές και το λέω και σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλήξουμε ευρωκειμένο το συντομότερων δυνατών. Πρόκειται για επίγον θέμα, για πολιτικό θέμα, το οποίο πρέπει να κλείσουμε το συντομότερο δυνατών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, ήδη είπε και ανέφερε ο συνάδελφος κύριος ε, Σεβερίν, η προσέγγιση της ε, δικής μας της ομάδας, η δική μας η στάση, ανέκαθεν ήταν μια στάση που έλεγε ότι ξεκινάμε από τις αρχές και όχι από οργανωτικής φύσεως θέματα. Τις αρχές που ανέφερε ο συνάδελφος, δηλαδή την διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, την απόδοση λόγου και όλα τα άλλα, αναμφίβολα αυτή η πρόταση αποτελεί μια απάντηση στην αναγκαιότητα να επιβεβαιωθούν οι αρχές. Εμείς λοιπόν ευχαριστούμε τους ε, εισηγητές ε, για τη δουλειά που μας ε, παρουσίασαν και για τη δουλειά που συνεχίζει να παρουσιάζεται, γιατί μας παρουσίασαν και μια τελευταία εκδοχή, η οποία περιλαμβάνει τις τελευταίες προτάσεις που διατυπώσαμε αναφέρομαι στις προτάσεις εκείνες που αφορούν στα θέματα του προϋπολογισμού του συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος θα υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για θέματα της ΚΕΠΑ, που νομίζω ότι είναι καθοριστικής φύσεως θέματα και το Κοινοβούλιο πρέπει ε, να εστιάσει την προσοχή του σε αυτά. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, είναι θέματα που βεβαίως και αφορούν την πραγματικότητα, ε, και ορισμένα εδάφια βεβαίως αφορούν αυτό που είπε ο κύριος Μπροκ, δηλαδή ένα σύστημα συνολικών ευρύτερων συμφωνιών που θα πρέπει να συμνοδεύουν την απόφαση του Συμβουλίου. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μπροκ. Δηλαδή πιστεύω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα από τα σημαντικότερα θέματα, γιατί εκεί θα μπορέσουμε να ε, εκφράσουμε την ε, πλήρη απόδοση λόγου της υπηρεσίας ε, απέναντι στο Κοινοβούλιο. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών προσπαθούμε να προσθέσουμε αυτά τα στοιχεία και ε, αναφέρομαι σε μια γνωμοδότηση δική μου στην Επιτροπή Προπολογισμών, όπου έκανα λόγο για ένα comprehensive document στα αγγλικά, δηλαδή ένα περιεκτικό έγγραφο περισσότερο από ένα ενοποιημένο ε, προϋπολογισμό, ο οποίος, ένα έγγραφο το οποίο θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε πολιτικά ε, τα διάφορα στοιχεία του προϋπολογισμού που αφορούν στην, ε, Επιτροπή, στην πολιτική εξωτερικής δράσης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν. Βεβαίως καθαρά τεχνικά αυτό που σας λέω δεν πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση. Κατά την άποψή μου, εξακολουθούν να υπάρχουν δύο προβλήματα όσον αφορά στη διατύπωση της πρότασης. Δηλαδή, στο κείμενο που μας μοιράστηκε, δεν υπάρχει αναφορά σε μία φράση που αφορά την πρόταση της κυρίας Άστον όπως αυτή τροποποιήθηκε από το τελευταίο Συμβούλιο, δηλαδή το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει πλήρης συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες γενικές διευθύνσεις ή απλά διευθύνσεις, όπως αναφέρεται στο έγγραφο Μπρόκ Φεχόφστατ. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το θέμα του συντονισμού είναι βεβαίως ένα θέμα το οποίο θετικά παρουσιάστηκε στην τελευταία εκδοχή της πρότασης της κυρίας Άστον μετά από τις συνεδρίες του Συμβουλίου, θεωρώ ότι αυτή η διατύπωση κυρίας Άστον πρέπει να διατηρηθεί, διότι ο συντονισμός σε, αυτή αυτήν την υπηρεσία είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο ενός μηχανισμού, ο ένας μηχανισμός ο οποίος έχει πλήρως υποέλεγχο το θέμα της ε, πολιτικής διαδικασίας και όχι μόνο το συντονισμό των υπηρεσιών και των εσωτερικών του δομών. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός συντονισμού πολιτικών, ο οποίος όμως δεν εξαντλεί το θέμα του συντονισμού ανάμεσα στις διάφορες διευθύνσεις ε, της ε, υπηρεσίας αυτής. Τη στιγμή μάλιστα που ο ε, Γενικός Διευθυντής είναι εκτελεστικό εκτελεστικό όργανο, υπάλληλος εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, όπως εξάλλου το ζητήσαμε και εμείς αυτό. Πρέπει ω εκ τούτου αυτό που σας είπα μόλι τώρα να διασφαλιστεί. Κατόπιν υπάρχει ένα πολύ πιο συγκεκριμένο θέμα και ενδιαφέρον το πώς θα επιληθεί, δηλαδή το θέμα του συντονισμού των ε, διαφόρων πολιτικών ε, που στις πολιτικές ε, που θα πρέπει να ακολουθούν. Κοιτάξτε, εδώ είναι αυτά τα θέματα που αφορούν στα στρατιωτικά και είναι σημαντικό να δούμε πώς ακριβώς θα ενταχθούν αυτές ε, οι πολιτικές, αν θα υπαχθούν σε αυτή τη διεύθυνση που θα αφορά στη διαχείριση των κρίσεων. Ένα άλλο θέμα κατά την άποψή μου, αφορά τα θέματα του προγραμματισμού. Κοιτάξτε, στον προγραμματισμό υπάρχει μια ε, συνεπέστατη λύση, η οποία συνδυάζεται με το πώς ε, θα λυθεί ένα καθαρά διοντολογικής φύσεως θέμα, δηλαδή η φύση αυτής της υπηρεσίας. Εγώ νομίζω ότι αυτό ε, θα έπρεπε να ενταχθεί καθαρά τεχνικά στην υπηρεσία προεπολογισμών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μην κολλήσουμε στις ε, λέξεις. Τη στιγμή, λοιπόν, που η υπηρεσία αυτή υπάγεται στην Κομισιόν, είναι σαφές, όπως λέει και ο κύριος Φεχόφστατ, ότι είναι πολύ πιο λογικό να οθήσουμε μέχρι το τέλος την αναζήτηση μιας φιλόδοξης λύσης. Δηλαδή, όλο τον προγραμματισμό να τον εντάξουμε σε αυτήν την υπηρεσία βεβαίως ανάλογα με τις ε, μεμονωμένες διευθύνσεις που αναφέρονται στην πρόταση. Αυτό που έχει σημασία και νομίζω αυτό το επενθύμισε και ο κύριος Βεχόφστατ είναι ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ε, αυτό το θέμα αντιμετώπισης διοντολογικής φύσεως ε, του ε, προβλήματος είναι λιγάκι διαφορετικό. Ε, πρέπει να πούμε ότι η πρόταση της κυρίας Άστον οδήγησε στο ότι οφείλουμε να αναδιατυπώσουμε αυτή την πρόταση για να υπάρχει ταύτιση με τον, ε, και με την υπηρεσία που θα καθορίζει το συντονισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κάπως κρίσιμο θέμα ε, που και σε σχέση με την πρόταση Μπρόκ φεχόφσετ αυτή η πολιτική καθοδήγηση και η σχετική πολιτική το, να το αναθέσουμε στην κυρία κυρία Άστον, ε, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά να υπάρχει και εμπλοκή του αρμόδιου επιτρόπου. Πρέπει να δούμε τώρα ποια είναι τα όρια ανάμεσα σε αυτήν την ε, ε, πολιτική καθοδήγηση και, τον, και την αρμόδια την είπα το εκπρόσωπο, είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει και σχέση με το γράμμα της συμφωνίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την αυτονομία αλλά και τις ε, πρόνοιες της ε, συμφωνίας, τα προνόμια όσον αφορά ε, τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη δική μας τη θέση, εμείς ε, βεβαίως ε, είμαστε πραγματιστές, όπως είπε και ο κύριος Σεβερίν. Εμάς μας ενδιαφέρει το πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε τις αρχές και λιγότερο τα τεχνικής φύσεως θέματα. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό το ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναδιατάξουμε και να αναδιατυπώσουμε αυτά τα θέματα ανάλογα με το πώς τελικά θα ε, εξελιχθεί η λύση που θα βρεθεί για το καθεστώς της υπηρεσίας. κύριε Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να δράξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Φεχόφστατ και τον κύριο Μπροκ, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια σειρά απόψεων ε, οι οποίες ε, τελικά ε, περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση μετά από τις εργασίες ε, που παρουσίασαν ο συντονιστή και ο σκιώδη συντονιστή. Ο κ. Σεβερίν έχει απόλυτο δίκιο που λέει ότι θα πρέπει οι εισηγητές άλλων επιτροπών που ασχολούνται με την υπηρεσία εξωτερική δράση, όλοι αυτοί να συνεργαστούν. Και αυτό αφορά κυρίως την Επιτροπή Προϋπολογισμών, Ελέγχου Προϋπολογισμών, αφορά την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, και την ε, Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Θέλω λοιπόν να εστιάσω την προσοχή μου σε δύο θέματα που αφορούν άμεσα την Επιτροπή των Συνταγματικών Υποθέσεων. Αναφέρομαι στον ε, μηχανισμό συντονισμού πολιτικών. Αυτό το μηχανισμό το θεωρώ πολύ σημαντικό, σημαντικό διότι Υπάρχει μια επιτροπή που λέει ότι τα θέματα, η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου, η επιτροπή αυτή λέει ότι τα, τα θέματα εξωτερικού εμπορίου δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με θέματα που εξετάζει η Επιτροπή Εξωτερική Δράση. Δεν έχουν καμία σχέση. Εγώ όμω θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε μια κοινή διατύπωση και ε, σε θέματα διαδικαστικά. Αυτό το βρίσκω σημαντικό. Και δεύτερον, αυτά για το περίφημο interfacing Νομίζω η διατύπωση που προτείνεται στο άρθρο 4.2 δεν αρκεί κατά την άποψή μου. Τουλάχιστον, όπως είπε και ο σήμερα, δεν νομίζω ότι αρκεί αυτή η διατύπωση για το περίφημο αυτό interfacing. Ε, νομίζω ότι πρέπει να το δουλέψουμε, δηλαδή να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό τον συνδυασμό των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και των άλλων που δεν την αφορούν. Πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το σημείο επαφής, αν θέλετε, αυτό το interfacing που ε, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν την εξωτερική πολιτική και να γνωρίζουν κατά πόσον πράγματι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να ελέγχει ε, για τους ε, τομεί ή στου τομεί, όπου έχουμε κάποιες αρμοδιότητες. Βεβαίω, δεν έχουμε αρμοδιότητες για όλους τους ε, τομεί. Αυτό πρέπει να το πούμε. Τελειώνοντας, όσον αφορά τον ε, προπολογισμό, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εδώ συμφωνώ με αυτά που είπαν οι προαλήσαντε κύριε Σεβερίν και Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να μην υψέλθω σε λεπτομέρειες. Ως αύκο θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ελπίζω ότι και οι άλλες επιτροπές θα ακολουθήσουν, θα ενστερνιστούν την πολιτική φιλοσοφία της έκθεσης. Πρόκειται για μια έξυπνη έκθεση θα έλεγα, αυτό συνεπεί που προσπαθεί να πετύχει το αδύνατο, την δηλαδή νέας δομής, που είναι μια ευρυδική μορφή από την σύλληψή της. Θέλω να χρησιμοποιήσουμε την κοινοτική ε, μέθο και αυτό το επιβραβεύω. Η προσπάθεια σημαίνει ότι θα συμμετάσχουν όλοι σε μια κοινή προσπάθεια και θα ήθελα να Στι τις οποίες τους ε, για το ότι προστατεύουν στο 7 ε, γάμα και στο 6, 6 την αρχή της γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητα. Ε, γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα σημαίνει ισχυρή υπηρεσία. Είναι αυτή η υπηρεσία θα απολαύει νομιμοποίησης και πολιτικής στήριξης ευρείας πολιτικής στήριξης και θα αντικατοπτρίζει άλλωστε και τους 700, τις των 727. Οι είναι αποφασισμένοι λοιπόν στον δρόμο αυτό. Πιστεύω ότι θα, είναι, θα σταθούν επάξια στην διαπραγμάτευση, την επικείμενη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο, κάτι το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή, ένα ερώτημα λέει ο Πρόεδρος. Ο Ήδη έθεσε το ερώτημα, αλλά το επαναλαμβάνω. Μπορείτε να μα πείτε λίγα λόγια σχετικά με την στάση του Συμβουλίου, γιατί πριν από έναν μήνα κάποια καθημερινή ξύπνησαν και συνειδητοποίησαν την πραγματικότητα. Συνειδητοποίησαν δηλαδή το θέμα της ε, συναπόφαση. Πώ πηγαίνει αυτή η διαπραγμάτευση. Φυσικά είναι και θέμα χρονισμού. Η δική μα θέση είναι ότι μπορούμε να κινηθούμε λίγο πιο αργά την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουμε το θέμα των Βρετανικών εκλογών, δηλαδή αν οι φιλελεύθεροι συνεχίσουν και πάρουν τις ψήφου που φαίνεται θα πάρουν, δεν ανησυχούμε, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την δική σας άποψη, ο κύριος Φερχόφστα. Δύσκολο να κάνω σχόλια για τις επικείμενες Βρετανικές εκλογές. Τι θα πω, θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία Υπάρχει βεβαίω η δυνατότητα να ζητήσουμε από του μετρούς να περιμένουν τι εκλογέ. Σε ό,τι αφορά το γενικότερο θέμα, θα ήθελα να ξεκινήσω με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Μπρόκ και εγώ επικοινωνήσαμε με τον κύριο Μωρατίνος... που εκπροσωπούσε την Ισπανική Προεδρία και η εντύπωση που μου δημιουργήθηκε είναι ότι αρχίζει να επιλαμβάνεται της κατάστασης η Ισπανική Προεδρία δηλαδή έχει σκοπό να συμβάλλει στο να προχωρήσει αυτό το, αυτός ο Ο κύριος Μπροκ και εγώ εξηγήσαμε στον κύριο Μορατίνος ποια είναι τα σημαντικά σημεία που αφορούν αυτή τη θέση και αρχίσαμε όχι μόνο να εξηγούμε τα συγκεκριμένα αυτά σημεία, το γνωρίζετε το πρόβλημα του προπολογισμού, το πρόβλημα των ε, αναπληρωτών, το πρόβλημα του συντονισμού και το πρόβλημα της συνοχής, της πολιτικής συνεργασίας και ανάπτυξης, που επίσης είναι ένα πρόβλημα ουσίας. Όλα αυτά τα θέματα συζητήθηκαν με την Ισπανική Προεδρία, με τον ε, κύριο Μορατίνο και σιγά σιγά άρχισαν, ε, άρχισαν να διαφαίνονται ορισμένες λύσεις. Πιστεύω ότι ο κύριος Μορατίνο μπορεί τώρα να ακούσει και τους, τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι στο Συμβούλιο και να αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν. Σε κάθε περίπτωση η Ισπανική Προεδρία θεωρεί ότι η συμφωνία που έγινε στο Συμβούλιο δεν σηματοδοτεί το τέλος της συζήτησης, αποτελεί φάση, βάση διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι κάτι που υπενθύμησε και το είπε και προς τα έξω η Ισπανική Προεδρία και είναι κάτι που επανελήφθηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε ο κύριος Μπρόκ και εγώ με την Προεδρία. Μπορώ να σας πω ότι περιμένουμε λίγο να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ισπανού Υπουργού Εξωτερικών τις επόμενες μέρες και τις επόμενες ώρες. Και αυτό σε ό,τι αφορά την άποψη του Κοινοβουλίου. Αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα της όλης διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, της πορείας των διαπραγματεύσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διάφορες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είμαι ευγνώμων προς όλα τα μέλη που πήραν το λόγο και που συνέβαλαν στη συζήτηση διατυπώνοντας προτάσεις. Θα προσπαθήσω να τις εξετάσω αυτές τις προτάσεις μία-μία και να τις σχολιάσω. Σε ό,τι αφορά το θέμα που έθεσε ο κύριος Σεβερίν για τον ενοποιημένο προπολογισμό, εγώ θα έλεγα να συμπεριληφθούν όλα στο τμήμα 3, όπως αναφέρεται στην τροπολογία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο όλα συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο μέρος του προπολογισμού. Το πρόβλημα αρχίζει όταν λέμε ότι θα δημιουργήσουμε μια ίδια υπηρεσία ε, σε ό,τι αφορά τις διοικητικές δαπάνες. Ε, οι λειτουργικές δαπάνες παραμένουν στο τμήμα 3. Το ένα βρίσκεται στο κεφάλαιο 5 και στο άλλο ε, στο 4. Ε, το να κάνουμε έναν ενοποιημένο προϋπολογισμό, βεβαίως εγώ είμαι νεοφερμένος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει μερικού κανόνε σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Έγινε μια διάκριση μεταξύ των διοικητικών και των ε, ε, ε, λειτουργικών δαπανών. Αυτό βεβαίω δεν σημαίνει ενοποιημένο προπολογισμό, γιατί γίνεται μια διάκριση υπάρχει μια όλη συζήτηση για τους special representatives. Πού θα πρέπει να του εντάξουμε αυτού διοικητικοί ή λειτουργικοί αν είναι ειδικοί εκπρόσωποι για ένα διάστημα πέντε ετών, είναι εύκολο να ενταχθούν στις διοικητικές δαπάνες. Όταν όμως πρόκειται για κάποιον που είναι συνδεδεμένος με μία συγκεκριμένη δράση, με μία συγκεκριμένη επιχείρηση, τότε μάλλον είναι λειτουργικό. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να αλλάξουν αυτοί οι κανόνες. Έχω την εντύπωση ότι μας χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να καταλήξουμε στον ε, υπάρχοντα προϋπολογισμό. Αλλά η λύση μας είναι η πλέον κατάλληλη, γιατί βάζοντας τα πάντα στο τμήμα 3 συμπεριλαμβάνονται και οι διοικητικές δαπάνες και οι λειτουργικές δαπάνες στο ίδιο μέρος ε, του προϋπολογισμού. Αυτά σε ό,τι αφορά το πρόβλημα αυτό ε, του ενοποιημένου προϋπολογισμού που έθιξε ο κύριος Σεβερίν. Τώρα, οι άλλες... Έγιναν και άλλες παρατηρήσεις. Να περάσω σε μερικές αυτές. Καταρχάς, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι ώστε ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων να είναι λειτουργικός. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το κείμενο ή τις ε, τροπολογίες. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό στην πρότασή μας. Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό κυρίως σε ό,τι αφορά το προσωπικό, τον προϋπολογισμό και το συντονισμό των πολιτικών. Σε επίπεδο πολιτικό βεβαίως έχουμε το μηχανισμό πολιτικής, σε πολιτικού συντονισμού για τον οποίο μιλήσαμε, αναφέραμε στις τροπολογίες. Αλλά ε, ε, εδώ μιλάμε για γενικό διευθυντή. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε το ρόλο του. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Από τη στιγμή που προβλέπεται αυτός ο ρόλος, ενδεχομένως θα μπορούσε να ενδυναμωθεί ε, έτσι ώστε όλη η διεύθυνση να μπορεί να συνεργάζεται υπό τη δική του καθοδήγηση, αφού αυτός θα είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Έγινε επίσης αναφορά στο θέμα της ανάπτυξης και της συνεργασίας. Αυτό αναφέρεται στο κείμενο. Αναφέρεται ότι σε ό,τι αφορά την πολιτική γυτνίας και την πολιτική ανάπτυξης είναι, ε, γίνεται αναφορά στο άρθρο 8. Έχουμε τροπολογία στο σημείο 2. Η εποπτεία, η άμεση, είναι άμεσης εποπτείας του, ε, άμεσης του Επιτρόπου προγραμματισμός είναι υπό την εποπτεία του ε, αρμόδιου επιτρόπου, όπως είναι και η εφαρμογή. Και αυτό υπό την εποπτεία του ε, αρμόδιου επιτρόπου. Συνεπώς, οι πέντε φάσεις του προγραμματισμού από το 1 μέχρι το 3 και το 4 και το 5 που αφορούν την εφαρμογή είναι υπό την άμεση εποπτεία, υπό την άμεση καθοδήγηση και ευθύνη του αρμόδιου Επιτρόπου για αυτό το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο υπέβαλα αυτές τις τροπολογίες για το άρθρο 8 παράγραφος 2. Βεβαίω, υπάρχουν συγκεκριμένες ε, προτάσεις που αφορούν μια διαφορετική διατύπωση που θα μας επιτρέψει να το καταστήσουμε αυτό περισσότερο σαφές. Πιστεύω όμως ότι το κείμενο ε, είναι αποδεκτό, δηλαδή ο Επίτροπος είναι αυτός που είναι υπεύθυνο. Αποτέλεσμα των τροπολογιών είναι ότι η πολιτική συνεργασία και ανάπτυξη καθώς και η πολιτική ηγετνία της, συνδέονται με την Επιτροπή, γιατί ο προγραμμισμός γίνεται από τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης και σε επίπεδο θεματικό και σε επίπεδο ε, γεωγραφικό που είναι συνδεδεμένες με την Επιτροπή. Κατά συνέπεια και ο προγραμματισμός είναι συνδεδεμένος με την ε, ε, Επιτροπή και τις αρμόδιες διευθύνσεις της. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθεί η υπάρχουσα κατάσταση. Θα μπορούσε κανείς να, να αποφασίσει για τον προγραμματισμό, αλλά θα μπορούσε να περιμένει ένα χρονικό διάστημα μέχρι τη στιγμή της ε, εφαρμογής. Αυτό βεβαίως είναι ένα πρόβλημα που δεν θα επιλύσουμε εδώ και σήμερα. Επίσης, ε, τέθη ένα θέμα για το interface. Στο άρθρο 4 προσπαθήσαμε να δώσουμε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Να περάσω στο κείμενο αγγλικά ένα τμήμα που θα είναι υπεύθυνο για το συντονισμό με τι αρμόδιε κοινοτικέ επιχειρήσει που θα αφορούν τι εξωτερικέ πτυχέ των εσωτερικών πολιτικών. Αυτό είναι το interface. Αυτό είναι ο ορισμό του interface. Αυτό που αποκαλούμε μία υπηρεσία στο εσωτερικό των ε, μιας άλλης που συγκεντρώνει όλες τις απόψεις που αφορούν το εξωτερικό εμπόριο, τις κλιματικές αλλαγές και όλα αυτά τα μεταφράζει, τα περνάει στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και εδώ οι δύο εισηγητές, αν υπάρχει μία άλλη διατύπωση που εξηγεί καλύτερα την ιδέα αυτή του interface, οι δύο συγητέ θα ήμασταν διατεθειμένοι να τη δεχτούμε. Κανένα πρόβλημα να καταβάλουμε μια προσπάθεια να επιφέρουμε βελτιώσει, διορθώσει στο κείμενο που αφορά το προβλεπόμενο interface, το άρθρο 4, παράγραφος 2. Thank you very much. We will have a special meeting in... Ευχαριστώ. Θα έχουμε μια ειδική συνάντηση στο Στρασβούργο για να συζητήσουμε το θέμα τη ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. ο Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Εγώ δεν θα αρχίσω να περισσότερο από ότι οι συναδελφοί μου. Νομίζω ότι γενικά είμαστε όλοι ικανοποιημένοι με τι προτάσει των εισηγητών, ούτω ή άλλω. Όμω, όμως, αν έτρεξα στη μνήμη μου και αν θυμάμαι καλά, στην Επιτροπή μα, αυτήν εδώ την Επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο, μιλούσαμε για ένα πιθανό ανώτατο όριο σε αυτό το όργανο και μιλούσαμε για το 5.000 και ξαφνικά ακούμε στο Συμβουλίο 8.000. Εάν το τρίτο προέρχεται από τα κρατημέλη, έχουμε 2.666, που είναι και συμβολικός αριθμός, προσωπικού δηλαδή που θα προέρχεται από τα κρατημέλη. 100 περίπου υπαλλήλοι από κάθε χώρα, ένα τέταρτο δηλαδή του προσωπικού του Εσθενικού Υπουργείου Εξωτερικών. Λίγο δύσκολο. Τέλο πάντων, θα μπορούσαμε τα ποσοστά, τα ποσοστά να παίξουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Ε, ε, εν πάση περιπτώσει η χρήσιμη πρόταση για τους διαπραγματευτέ θα ήταν να υπενθυμίσουμε στον κύριο Μαρατίνο ότι στην συζήτηση περικροπολισμού το κοινοβούλιο αυτό ε, δεν θα δώσει μάχη υπέρ του 5.000. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως, ενδεχομένως να δεχθούμε και το 8.000. Δεν ναι, μου φαίνεται καλό ως στόχος. Ε, βλέπω τώρα ότι η συζήτηση θα περάσει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα τα πούμε αυτά στις 22 Μαου. Ευχαριστώ. Και να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Πρόσβαση σε έγγραφα. Πρόσβαση τεκμηρίωση, ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο οπω όλοι γνωρίζετε έχει παγώσει για χρονικό διάστημα. Περιμέναμε την νέα Κομισιόν. Η Επιτροπή έχει συζητήσει το θέμα και βέβαια και δικό μας ε, θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού. Οπότε δίνω αμέσω τον λόγο στον εισηγητή, στην κυρία Γιάννη Uudistettu Ο κανονισμός αυτός ε, που αφορά στη δημοσίευση των εγγράφων ε, έχει ήδη διάρκεια ζωής ε, δύο ετών και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έχει και ο τέλος. Πέρυσι ε, την Άνοιξη διακόπηκαν οι διαβουλεύσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το επιθυμούσε και η συγγήτρια. Το φθινόπωρο ξανάρχισαν και το Δεκέμβρη το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα. Το Κοινοβούλιο λοιπόν στο ψήφισμα αυτό καλεί την Κομισιόν να καταθέσει μια νέα πρόταση, όμως ε, τελικά δεν έγινε τίποτα. Η Κομισιόν ε, αρνήθηκε ε, διότι υπήρχαν, ε, υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα στην Κομισιόν και το Συμβούλιο. Και τώρα πρέπει κάπως ε, να προχωρήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να αναφερθώ στις ε, διάφορες απόψεις, αλλά θα μου επιτρέπετε, επιτρέψετε να ξεκινήσω με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή η συνθήκη της Λισαβόνας. Τροποποιεί την ε, νομοθετική βάση του κανονισμού με την εξή έννοια, ότι κατά το παρελθόν ο κανονισμός ο οποίος ε, ήδη εξετάστηκε πριν από δύο χρόνια, ο κανονισμός ε, αυτός ένωσε τότε το Συμβούλιο, την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και τώρα μετά τη θέση ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας ο κανονισμός ε, αυτός αφορά και το Συμβούλιο, την Europol, ε, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, εδώ πρόκειται για μία επέκταση της ισχύω του κανονισμού. Να πω και κάτι άλλο που και αυτό έχει σχέση με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Πιστεύω ότι πολύ εξημών υποστηρίξαμε τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας, γιατί ε, πιστεύαμε ότι θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός λοιπόν ο κανονισμός που κατέθεσε η Κομισιόν, αν δούμε λιγάκι τα μεμονωμένα άρθρα του κανονισμού, θέλω να σας πω ότι δεν διαπιστώνουμε ενίσχυση της διαφάνειας. Εκτός από το ότι αυξάνεται ο αριθμός ε, των άμεσα αρμόδιων οργάνων, δηλαδή αρμόδια, ε, δεν είναι πλέον μόνο τα όργανα Κομισιόν και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και άλλα. Πάντως, άμεση ενίσχυση της διαφάνειας εμείς τουλάχιστον δεν διαπιστώνουμε. Τώρα, όσον αφορά τα μεμονωμένα άρθρα, ο κανονισμός ε, της έννοιας έγγραφο και πώς ε, καταχωρίζουμε τα διάφορα έγγραφα. Τόσο στην πρόταση της Κομισιόν, όσο και στην πρόταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, υπάρχει ένα ε, πολυδιάστατο σύστημα ταξινόμησης. Η ταξινόμηση γίνεται ανάλογα με το κατά πόσον ε, τα έγγραφα είναι δημόσια ή διαβαθμισμένα. Και επ' αυτού υπάρχει διάσταση απόψεων. Όσον αφορά γενικά τον ε, ορισμό, δεν έχουμε τίποτα να πούμε, αλλά την ε, ε, ταξινόμηση και καταχώρηση των εγγράφων σε διάφορες κατηγορίες ε, διαβάθμισης, αυτό ε, δημιουργεί προβλήματα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, αυτή η καταχώρηση αφορά την εργασία, στα έγγραφα που αφορούν τους δύο θεσμούς και όχι στα έγγραφα που είναι προσπελάσιμα για τους πολίτες. Το Δεκέμβριο στο ψήφισμα του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε από το σύνολο των βουλευτών, εκεί εμείς ε, λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ε, σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στη δυνατότητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στο έγγραφο και ανάμεσα στα έγγραφα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους ε, δύο θεσμούς, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους θεσμούς είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα όμως, αυτό είχαμε πει τότε, τώρα τι γίνεται, κάπως μπερδεύονται πάλι τα πράγματα. Ως εκ τούτου, αντί να έχουμε μεγαλύτερη, έχουμε λιγότερη διαφάνεια. Μπορώ βέβαια να δώσω και ε, μια καλή αιτιολόγηση για αυτόν τον τρόπο καταχώρησης εγγράφων. με την έννοια ότι αυτή η καταχώρηση των εγγράφων βασίζεται στη διαβάθμιση που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως υπάρχει ένας κανονισμός του 2001 όπου σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό το όλο θέμα ρυθμίζεται στο πλαίσιο μιας διαθεσμικής συμφωνίας και εκεί ακριβώς αναφέρεται και η δυνατότητα πρόσβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διαβαθμισμένα έγγραφα. Ε, θέλω να πω και κάτι άλλο. Τίθεται το θέμα κατά πόσον ε, τα κράτη-μέλη έχουν ε, το δικαίωμα της αρνησικυρίας, τουλάχιστον όσον αφορά τα δικά τους έγγραφα. Αυτή η πρόταση κατά κάποιον τρόπο προβλέπει το δικαίωμα της ε, αρνησικυρίας. Η πρόταση της ε, Κομισιόν δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ασκήσουν το δικαίωμα της ε, αρνησικυρίας, να απαγορέψουν την ε, πρόσβαση στα δικά τους έγγραφα. Άρα δηλαδή σαφώς αυτό είναι δικαίωμα βέτο των ε, κρατών μελών. Εμείς όμως δεν συμφωνούμε με αυτό. Θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν κοινοί κανόνες και όχι κανόνες όπου το κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει μόνο του. Αυτά, αν θέλετε, είναι τα δύο ε, θέματα όπου υπάρχει η πιο έντονη διάσταση απόψεων. Δηλαδή, ε, καταχώρηση και ε, ορισμός των εγγράφων, ε, καταχώρηση με βάση τη διαβάθμιση, το βαθμό διαβάθμισης και κατόπιν και πρόσβαση στα έγγραφα των κρατών μελών. Υπάρχουν και κάποια άλλα, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικότερα. Ε, κυρίως όσον αφορά την ε, πρόσβαση στα έγγραφα κρατών μελών, εκεί σας είπα δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, διαφοροποιημένες ρυθμίσεις. Η πρόταση Κομισιόν έχει κατατεθεί και αυτό που επικρίνει και η πρόταση πολιτικών ελευθεριών είναι ότι όλα αυτά όμως ε, δεν ε, συμβαδίζουν με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ελήφθη τον περασμένο Δεκέμβρη. Αυτή ήταν τότε η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουμε αυτό που αποφασίσαμε το Δεκέμβρη. Όμως και πάλι να σας πω ότι εγώ είμαι στη διάθεσή σας να εγκρίνω και άλλες ε, απόψεις γιατί είναι πολύ περίπλοκο θέμα και επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Ε, αποκινούμε την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα έπρεπε ή προβλεπόταν να υπάρξει μία ακρόαση τον Ιούλιο, που δεν θα γίνει όμως. Βέβαια θα ήταν απαραίτητο να λάβει η χώρα μια τέτοια ακρόση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα περίπλοκο θέμα και πρέπει όλοι από κοινού να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. The floor is open. Señor favor. Muchas gracias, señor presidente. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η χθεσινή συζήτηση σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ή μάλλον συμφωνήσαμε όλοι ότι σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση υπάρχει μια πολιτική βάση και είναι σημαντικό να υπάρχει μια ενιαία βάση. Έγινε αναφορά ότι θα πρέπει να τονίσουμε το θέμα της ύπαρξης ενός ευρωπαϊκού λαού. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα, αλλά στις αποφάσεις, αλλά και σε όλες τις διαδικασίες, σε όλα τα έγγραφα που οδήγησαν στην υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης απόφασης. Από το 2001 έχει καταγραφεί μεγάλη πρόοδος. Οι πολίτες, δηλαδή οι λαοί της Ευρώπης έχουν τα μέσα για να μπορούν να παρεμβαίνουν στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λογικό, συνεπώς, το ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος και σε σχέση με όσα αποφασίστηκαν το 2001 για τη διαφάνεια στην πρόσβαση στα έγγραφα. Η απόφαση αυτή για μια μεγαλύτερη διαφάνεια είναι κάτι που συναντάμε όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε πολλές χώρες από το 2000 μέχρι το 2010 ενέκριναν νόμους που δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα έγγραφα. Σε ορισμένες χώρες, μιλάω για την Ισπανία, μια χώρα που γνωρίζω, επανεξετάζεται η νομοθεσία σχετικά με αυτό το θέμα και αυτή η αναθεώρηση έχει στόχο να δώσει περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες για πρόσβαση και για μεγαλύτερη τεκμηρίωση. Αυτό σε ό,τι αφορά τα έγγραφα που οδηγούν σε μια δεύτερη φάση στη λήψη μιας απόφασης. Δεν θα ήταν σκόπιμο να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Έχουμε έναν κανονισμό, ο οποίος εφαρμόστηκε μέχρι τώρα αρκετά καλά έχει όμως εγκρίθηκε πριν από 10 χρόνια. Θα ήταν σκόπιμο λοιπόν να τον επανεξετάσουμε. Σε μία προηγούμενη συνεδρίαση θα ήθελα να θυμίσω ότι η Επιτροπή εξέφρασε μία συντηρητική θα έλεγα θέση. Ήταν κατά της ιδέας του να γίνουν δεκτές ε, νε... αλλαγές. Η άποψή της ήταν ότι το σύστημα είναι λειτουργικό και δεν υπάρχει λόγος αλλαγής του. Θα ήθελα να θυμίσω ότι πήρε το λόγο ο κύριος Νταφ για να πει ότι αυτή είναι η καινούργια επιτροπή. Αυτό όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα μέλη, μιλάμε για την εκτελεστική επιτροπή εδώ, αλλά γιατί ήταν αποτέλεσμα μιας θεσμικής μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν σημαντικό να καταλάβουμε εάν η νέα επιτροπή θα επιθυμούσε να δώσει περισσότερα μέσα, να ε, θέσει ε, περισσότερα μέσα στη διάθεση των πολιτών για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα. Προσέθεσα και εγώ με τη σειρά μου ότι η Επιτροπή αντέδρασε όπως ήταν αναμενόμενο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε θεσμικές σχέσεις υψηλού επίπεδου με την Επιτροπή για να μπορέσουμε να δούμε αν θα ήταν διατεθειμένη να δεχτεί ορισμένες τροποποιήσεις, ε, τροπολογίες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Και εγώ, όπως έλεγε και η συγγήτρια, είμαι της άποψης ότι δεν είναι λογικό σε ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει πρόσβαση κατά 100% και σε άλλες χώρες πρόσβαση κατά 35%. Πιστεύω ότι είναι λογικό να λάβουμε υπόψη μας ορισμένες εθνικές ιδιαιτερότητες. Όχι σε ό,τι αφορά το γενικό κατόφλι που προβλέπεται για την πρόσβαση των πολιτών. Θα πρότεινα συνεπώ οι εισηγητές των Επιτροπών ΛΥΜΠΕ και ΑΦΚΟ να εξετάσουν την διοργάνωση μια συνάντηση υψηλού επίπεδου με του υπεύθυνους τη Επιτροπή ή να εξετάσουν κατά πόσον κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης θα ήταν δυνατόν να θέσουμε ορισμένες ερωτήσεις σε ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και να δούμε εάν θα ήταν διατεθειμένη να διευρύνει την πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις. come back to the question. Θα παρέλθουμε στην ακρόαση με τους συντονιστές, γιατί το αίτημα είναι η ακρόαση είναι κοινή και από τις δύο επιτροπές, οπότε θα το ξαναδούμε αυτό. Άλλος που θέλει το λόγο, για κάποιο άλλο θέμα ενδεχομένω εισηγητρία. Να πω μόνο ότι συνάντησα τον Επιτροπό την, στο περασμένο Στρασβούργο και ζήτησαμε το θέμα και μάλιστα συμφωνήσαμε ότι πρέπει να βρούμε λύση. Έχουν περάσει δύο χρόνια. Ήρθε η ώρα και δυστυχώς έχουμε ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι συμφωνίε πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επίτροπή, Πολ Ράζελ είναι ο εισήγητη. Πολ παρακαλώ. Πρώτα ευχαριστώ. Από την περασμένη μας συνεδρίαση τότε δηλαδή που μιλήσαμε για το θέμα αυτό. Δεν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Υπενθυμίζω πάντως τι έχουμε κυρίως πετύχει ως τώρα και τα τρία τέσσερα εκκρεμή θέματα στη σύντηση μας με την Κομισιόν. Μετά το ψήφισμα της 9ης Φεβρουαρίου καταφέραμε, πρέπει να πω, να θεσπίσουμε νέους κανόνες για την συμμετοχή επιτρόπων σε εκλογικές, προεκλογικές εκστρατείες. Επίσης θέσαμε συγκεκριμένες διατάξεις στον επαναρτημά όσον αφορά την ενημέρωση προς το Κοινοβούλιο για τι αντίστοιχε τη Κομισιόν με Εθνικού Συμπειρογνωμόνε για την προετοιμασία και εφαρμογή κοινοτική νομοθεσία, ακόμη και το λεγόμενο soft law. το πετύχαμε τι περασμένε εβδομάδε. Γιατί οι συναντήσει με του Εθνικού Συμπειρογνωμόνε και το soft law ήταν ε, θέματα τα οποία μα δυσκόλυψαν πολύ. Έχουμε επίση διατάξει όσον αφορά την συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και τη Κομισιόν στον τομέα των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια συμπεριλαμβάνει νομοθεσία σχετικά με τι αιτιολογημένε γνώμες. Η σχέση λοιπόν με τα εθνικά κοινοβούλια, ένα θέμα το οποίο έκλεισε, ήταν σημαντικό θέμα πρέπει να πω. Σημειώθηκαν επίση βελτιώσει στην διαδικασία τη περιπτώσει που το Κοινοβουλίο γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Βελτιώθηκε εκεί η σχετική διαδικασία και αυτό ήταν ένα ενδιαφέρον σημείο. και έχουμε επίση και κάποιους κανόνες για την επιβεβαίωση των κατευθυντηρίων γραμμών περιορισμένων θεμάτων για να λαμβάνετε καλύτερη υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου. Αυτά είναι για το μέλλον, πάντως, και αφορούν, επαναλαμβάνω, την ε, έγκριση της επόμενης Επιτροπής, της επόμενης Κομισιόν. Θα συνεχίσουμε να συζητούμε μέχρι το επόμενο Στρασβούργο. Πρέπει έως τότε να καταλήξουμε σε συμφωνία επί πολύ δύσκολων ζητημάτων. Το ένα είναι η αναθεώρηση των σημερινών του πιστεμένων διατάξεων όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των εγγράφων, κάτι το οποίο σχετίζεται με το, με το οποίο μόλις συζητήσαμε. Έλεγα λοιπόν για την εμπιστευτικότητα των εγγράφων. Οι σχετικές διατάξεις πρέπει να αναθεωρηθούν Θυμίζω επίση ότι δύσκολα καταλήξαμε σε συμφωνία όσον αφορά τις λεπτομερείς διατάξεις για τον προγραμματισμό δηλαδή το Κοινοβουλίο Κομισιόν πριν εγκριθεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, να έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Αυτό δεν ήταν και δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή να υπάρχει ένα κοινό κείμενο επί αυτών των ζητημάτων. Δηλαδή το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Φυσικά θα επιθυμούσαμε να έχουμε με προξάρχουσα θέση ω κοινοβούλιο στον καθορισμό του ετησίου προγράμματος εργασιών. Αυτό όμω είναι δύσκολο. Οπότε θα έλεγα ότι το πιο λεπτό ζήτημα και αυτό το οποίο μας δυσκολεύει είναι οι διεθνείς διαπραγματεύσεις. Οι λεπτομερείς δηλαδή διατάξεις σχετικά με τον ενισχυμένο ρόλο του Κοινοβουλίου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Ίσως βάσει και ενός νέου παραρτήματος και με βάση βεβαίως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά και πάλι είναι δύσκολα. Η θέση θα λέει, της Κομισιόν δεν είναι και αυτή εύκολη, διότι η Κομισιόν καταρχήν δεν ήθελε να θεσπίσει συγκεκριμένε διατάξει στο πλαίσιο αυτή τη συμφωνία πλαίσιο, διότι θεωρεί ότι το θέμα αυτό πρέπει να ρυθμιστεί επευθείας με τον αρμόδιο αντιπρόσωπο που είναι αρμόδιος για τις εξωτερικές ε, σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφαλεία κλπ. Αυτό το θέμα έχουμε λοιπόν στις εξωτερικές σχέσεις. Εμείς προσπαθούμε καταρχήν να συμφωνήσουμε με κάποιο κανόνα βάσει του οποίου τα μέλη του Κοινοβουλίου θα μπορούν να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο, έστω και ως παρατηρητέ του ΣΥΠΗΝ, ω μόνιμοι παρατηρητέ αν θέλετε, στι διεθνείς αυτέ διαπραγματεύσει. Όμω, εδώ δεν έχουμε μόνο την Κομισιόν. Έχουμε μια ειδική θεσμική θέση του Αντιπροέδρου Αρμοδίου για τις εξωτερικές σχέσεις και του είπα το πρόσωπο το, να τα συγκεράσουμε όλα αυτά ήταν πολύ δύσκολο. Συνοψίζω, τρία είναι τα εκκρεμή θέματα. και στην καρδιά φυσικά της διαπραγματευσή. Το πρώτο είναι η εμπιστευτικότητα των εγγράφων. Το δεύτερο είναι το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν. Και τρίτον, ο ρόλος του Κοινοβουλίου στον σχεδιασμό, στην κατάσταση του ετησίου προγράμματο. Και τέλο, εξίσου σημαντικό, θα λέγαμε μάλιστα ότι είναι και το πιο δύσκολο θέμα, είναι οι διεθνεί διαπραγματεύσει και ο βαθμό συμμετοχή, το επίπεδο συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτέ. Αυτά είναι τα τρία κυρία ζητήματα που συνεχίζουν να εκκρεμούν και από των οποία δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, Άντριου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Όντω δεν έχει σημειωθεί και κάποια σπουδαία πρόοδο. Πάντω έχει σημασία η επισπέυδουσα ομάδα, το steering group ε, που συστήθηκε να προσπαθήσει να βελτιώσει μεταξύ άλλων και τα τη συνεργασία μεταξύ ημών και των Εθνικών Κοινοβουλίων στο πλαίσιο τη ε, συμφωνία πλαίσιο. Αυτό πρέπει να συστήθει και να κλείσει με την Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν έχει ρόλο να διαδραματίσει στην βελτίωση της ποιότητας της διακοινοβουλευτικής εργασίας Και τέλος, ένα άλλο θέμα το οποίο μάλλον υποτιμήσαμε. Βάσει τη συνθήκη υπάρχει υποχρέωση για τα τρία όργανα Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Κομισιόν να συμφωνούν βεβαίως επί ενός πολιτούς προγραμματός εργασιών για πέντε συγκεκριμένα έτη. Αυτό είναι ουσιώδες για την απόδοση και η αποτελεσματικότητα και συνέχεια της νομοθετικής και πολιτικής μας εργασίας. Διότι αν αποτύχουμε προκειμένου τα προγράμματα προεδριών θα συνεχίσουν να λειτουργούν αποσπασματικά. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να περιγράψουμε αυτή τη δυσκολία είναι να καταστρώνονται αυτό συνεπεί πενταετή προγράμματα με τα οποία θα συμφωνούν και τα τρία θεσμικά όργανα. Κατανοώ το πρόβλημα για τα αιτήσια προγράμματα Εκεί πάλι υπάρχει ένα πρόβλημα λόγω και μόνο των καθυστερήσεων που παρουσιάζονται σε αιτήσια βάση και προκειμένου φέτος ε, λόγω των καθυστερήσεων με την Κομισιόν. Έχετε συζητήσει καθόλου το θέμα λοιπόν των πολιετών προγραμμάτων, αυτήν την ερώτησή μου. Άλλο. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι δεν συζητήσαμε αυτό το πρόγραμμα, το πρόβλημα του πολιετού προγράμματος. Συζητήσαμε όμως την ανάγκη για μια διαθεσμική συμφωνία που να έχει μια τρισδιάστατη συμφωνία μια συμφωνία όπου η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορούν να έχουν μια κοινή βάση διαλόγου. Συζητήσαμε το θέμα με την Επιτροπή, και το, αλλά και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν την άποψη ότι το Συμβούλιο δεν έχει τόσο ανοιχτή στάση. Δεν προσφέρεται τόσο πολύ για μια ευρεία διαθεσμική συμφωνία. Υπάρχουν, θα έλεγα, μερικές επιφυλάξεις, μερικές δυσκολίες το να γίνει δεκτή μια ευρεία τριμερής συμφωνία. Βεβαίως, θα επικοινωνήσουμε με το Συμβούλιο, αλλά όχι στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Η εντολή της ομάδας εργασίας για αυτή τη συμφωνία πλαίσιο είναι συγκεκριμένη, αφορά αυτό και μόνο τη συμφωνία μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Μερικές φορές η Επιτροπή μας στέλνει απαντήσεις όπου αναφέρει ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν επί ενός ή άλλου θέματος, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Πιστεύω λοιπόν ότι ενδεχομένως και θα έλεγα ότι αυτή είναι η άποψη του Προέδρου αυτής της ομάδας εργασίας και ξέρετε ότι ε, ε, αναφέρομαι στον κύριο Λένα από κοινού με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου προσπαθεί να εδραιώσει μια θέση με το, σχέση με το Συμβούλιο. Πιστεύω ότι τώρα αυτό είναι πιο εύκολο, γιατί υπάρχει ένας πρόεδρος του Συμβουλίου με συγκεκριμένη ε, θητεία 2,5 ετών. Συνεπώς, ε, θα είναι ενδεχομένω πιο εύκολο να επιτευχθεί μια συμφωνία, ένα είδος θεσμική συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου αλλά το πολιετές πρόγραμμα θα έλεγα ότι δεν είναι ένα θέμα που συζητήσαμε στην ομάδα εργασίας που ασχολείται με αυτή τη συμφωνία πλαίσιο. Anyone else? Κάποιος άλλος, κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Ωραία. Περνάμε λοιπόν το επόμενο και τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης, εκλογές του Κοινοβουλίου, ο Άντριο Νταφ ήταν εισηγητή στο προηγούμενο Κοινοβούλιο και συνεχίζει το έργο του. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε νομοθετική πρωτοβουλία και νομίζω ότι μας αφορά ιδιαίτερα το θέμα ως βουλευτές. Δίχως καθυστέρηση λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντάφιν. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που δίνετε ευκαιρία να υποβάλω αυτή την έκθεση. Δεν υπάρχουν πολλοί παρόντες και το μόνο που ελπίζω είναι να μην αποτελεί ένδειξη της αδιαφορίας του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την ε, εικόνα που δίνει προς το εκλογικό σώμα. Δαπανίσαμε χρόνο για να αλλάξουμε τις συμφωνίες και το βασικό αποτέλεσμα είναι ότι αυξήθηκαν οι εξουσίες του Κοινοβουλίου. Η σύνθεση του Κοινοβουλίου τέθηκε στο περιθώριο αυτής της παρατεταμένης διαδικασίας και νομίζω ότι ήρθε πλέον η ώρα για να ασχοληθούμε και πάλι με αυτά τα θέματα. Θέματα νομιμότητας, θέματα του κατά πόσον είναι δημοφιλές το κοινοβούλιο ή τις εικόνες που προβάλλει το κοινοβούλιο προς τα έξω είναι πολύ σημαντικά. Και είναι πολιτικό μας καθήκον να ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά με έναν επικοδομητικό και προοδευτικό τρόπο. Όπως ανέφερε ήδη ο πρόεδρος, ο τομέας είναι ένας τομέας επί το οποίου το Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλλει στο να γίνουν αλλαγές. Ε, Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε την εκλογική διαδικασία. Έχουμε τη δυνατότητα και την εξουσία να προτείνουμε αλλαγές στη σύνθεση του Κοινοβουλίου και έχουμε και την εξουσία να προτείνουμε αλλαγές στις συνθήκες. Όλες αυτές οι εξουσίες αναφέρονται σε αυτή την έκθεση που σας υποβάλλουμε. Αν θα μπορούσα να περιγράψω, ή αν θα μπορούσα να αναφερθώ στα έγγραφα αυτά, θα έλεγα ότι είναι μάλλον πολύπλοκα. Το πρώτο είναι μία έκθεση του Κοινοβουλίου. Το δεύτερο είναι το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που θα αλλάξει το τα, τα όσα προβλέθησαν το 1976 καθώς και τις προτινόμενες τροπολογίες σε αυτή την πράξη. Το τρίτο έγγραφο που συμπεριλαμβάνεται το φάκελο είναι ο νόμος του 76 ο οποίος αναθεωρήθηκε τρεις φορές, αν δεν κάνω λάθος, από το 1976, αλλά που δεν έχει δημοσιευθεί που άλλου. Είναι μάλλον περίεργο ότι η επίσημη εφημερίδα των κοινοτήτων δεν κατάφερε να δημοσιεύσει μία ε, νοποιημένη εκδοχή του. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να αναφερθούμε στην επικαιροποιημένη εκδοχή. Το τέταρτο έγγραφο που διανεμήθηκε σήμερα είναι μια επεξηγηματική δήλωση. Είναι εκτενής και δεν έχει μεταφραστεί ακόμα από τα αγγλικά σε κάθε περίπτωση βρίσκεται σε φάση μετάφρασης. Εδώ γίνεται μια ιστορική περιγραφή της όλης έννοιας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, της εκλογής του Κοινοβουλίου και των αλλαγών, των συνθηκών που επηρέασαν την διαδικασία και τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήσαμε από τις εκλογικές εκστρατείες και που θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε τις διαδικασίες και κατά πόσο τα κατάφεραν να κινήσουν τον ενδιαφέρον και να δυναμώσουν την αντιπροσωπευτική την δυνατότητα αντιπροσώπευσης του έχει το Κοινοβούλιο. Και καταλήγει στο τέλος ορισμένα συμπεράσματα. Συμπεράσματα που προσπάθησα να αναφέρω στην έκθεσή μου. που βρίσκονται στην αρχή του φακέλου. Η επεξηγηματική δήλωση έχει πέντε παρατήματα και θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα σε αυτά. Το πρώτο αφορά την έκθεση Αναστασόπουλου που ενέκρινε το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 1998 νομίζω Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλαμε να επιλύσουμε αυτά τα πολύπλοκα θέματα. Έχει περάσει πολύς χρόνος και θεώρησα ότι ήταν αναγκαίο να φρεσκάρουμε λίγο τη συλλογική μας μνήμης σε ό,τι αφορά τον τρόπο που βλέπαμε τα πράγματα τότε. Βεβαίως πριν από την υπογραφή της συνθήκης της Νίκαιας Το δεύτερο παράρτημα στο επεξηγηματικό μνημόνιο, που είναι σελίδα 24, είναι ένας χάρτης που αναφέρεται στην κατανομή των εδρών. δυστυχώς δεν γίνεται μία αναφορά στις περιπτώσεις ε, της φθήνουσας αναλογικότητας ε, και που δεν επιτυγχάνεται. Εάν ε, κοιτάξετε από κοντά αυτό το κατάλογο, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι στο παρόν κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο των 736 εδρών, υπάρχουν εννέα χώρες που δεν κατάφεραν να σεβαστούν την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Και ακόμα και αν προσθέσουμε τις 18 έδρες από τον οποίο θα αποφασίσουμε την πέμπτη, δηλαδή αν θα εγκριθούν ή όχι, αν προσθέσουμε και τις 18 έδρες, υπάρχουν 5 χώρες που δεν συμμορφώθηκαν με αυτή την αρχή. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα από όλα αυτά ότι η πολιτική επηρεάζει την κατανομή των εδρών και νομίζω ότι η μέθοδος που ακολουθήσαμε στο παρελθόν δεν είναι μια μέθοδος αποτελεσματική για την διανομή και την κατανομή των εδρών. Ναι. Και πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε αυτή την φόρμουλα. Όπως διαπιστώνετε σε αυτό τον χάρτη που σας υπέβαλα, το διάγραμμα, έχω βάλει την εναλλακτική πρόταση του 2014. Νομίζω ότι τότε θα, θα πρέπει να επιληφθούν, ε, επιληφθεί η κορατή Ισλανδία. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλό, καλή πρόταση, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι η μόνη που σέβεται την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Συνεπώς, είναι μια βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με την παρούσα και είναι σύμφωνη και με τις συνθήκες. Θα πρέπει όμως να το δούμε στα πλαίσια της συμφωνίας, γιατί υπάρχει η μείωση του πληθυσμού στη Γερμανία, στη Γαλλία και η Βρετανία. Στη Γαλλία και η Βρετανία αυξάνεται ο πληθυσμός και αν η Γερμανία επιμείνει στον αριθμό των βουλευτών που είχε το 96, θα πρέπει να αντισταθμίσουμε τις, ε, τους Γάλλους και τους Βρετανούς με μια σημαντική αύξηση. Α. Έχουμε, έχουμε τους Έλληνες, τους Ολλανδούς, ε, ε τους Βέλγους που θα, θα δούμε συμπιέζεται ο αριθμός των βουλευτών. Παρόλα τα οικονομικά προβλήματα αυτών των χωρών, πρέπει να δούμε αν θα ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν μία μείωση της εκπροσώπησής τους στο Κοινοβούλιο. Θα δείτε στην γραφική παράσταση που είναι στη σελίδα 25 του επεξεργηματικού αυτού μνημονίου Βέβαια είναι δύσκολο να τα καταλάβετε έτσι όπως είναι ασπρόμαυρα, αλλά η πιο μαύρη από τις ε, ε, γραμμές, τις στήλες είναι η παρούσα κατανομή και μετά βλέπετε τα ανώτατα και εκατότατα σημεία που δείχνουν την φθήνουσα αναλογικότητα. Ενώ η θεά, η γκρι περιοχή είναι μία παραβολή, όχι ακριβώς παραβολή, είναι κάτι συναφές με μια παραβολή που εξηγεί την εναλλακτική λύση που υπέβαλα τον Ιούλιο του 2014. Συνεπάγεται μία βελτίωση, όχι βέβαια την επίτευξη της τελειότητας. Βασίστηκα βεβαίως στον παρόντα πληθυσμό όπως δημοσιεύτηκαν από την Eurostat πέρσι το φθινόπωρο το 2014. Βεβαίως θα έχουν έρθει σημαντικές αλλαγές στον πληθυσμό. Ο πληθυσμός της κάθε χώρας αλλάζει και θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτή η αυξομοίωση του πληθυσμού. Αν περάσουμε σε σελίδα 26, θα δείτε μια γραφική παράσταση που μάλλον θα μας θλίψει. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την προσέλευση στις εκλογές του Κοινοβουλίου από το 1979 και μετά. Όπως γνωρίζετε αυτή η προσέλευση συγκαλύπτει εσωτερικές διακοιμάσεις. Παρόλα αυτά, είναι μια ιδιαίτερα αλγινή εικόνα για όλους εμάς εδώ, που μάλλον πιστεύουμε στην έννοια της διακρατικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Στη σελίδα 27 βλέπετε μία γραφική παράσταση που αφορά τα δύο φύλλα, την εκπροσώπηση των δύο φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έλεγα ότι προσεγγίζουμε ένα σημείο που θα υπάρχει ίση εκπροσώπηση, αλλά θα πρέπει να δούμε πόσο απέχουμε ακριβώς. Ο τελευταίος πίνακας, το παράρτημα 5, προσπαθεί εν συντομία να περιγράψει τις 27 εκλογικές διαδικασίες για το Κοινοβούλιο. Ελπίζω να είναι ακριβής αυτός ο πίνακας. Αν οι συνάδελφοι θεωρούν ότι δεν έχω συμπεριλάβει τις πολύπλοκες εθνικές εκλογικές τους διαδικασίες, θα ήμουν ευγνώμων αν μου το ανέφεραν. Αυτή, λοιπόν, ήταν μια περιγραφή των εγγράφων που έχετε μπροστά σας. Θα ήθελα τώρα, εν συντομία, να περιγράψω τις προτάσεις που υποβάλλω. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα μέχρι το 2014 να έχουμε κλείσει τα πάντα. Έχουμε χρόνο βέβαια, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Ε, θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε να ε, διαβουλευόμεθα με τα πολιτικά κόμματα, γιατί πρέπει να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, αλλά και η ΜΚΟ, η Επιτροπή, αλλά και το Συμβούλιο καλούνται να τοποθετηθούν και ελπίζω ότι ε, στο τέλος θα έχουμε και λίγο χρόνο να μιλήσουμε για το την κατάλληλη χρονική στιγμή, τον χρονισμό της όλης αυτής ε, διαδικασίας. Στόχος λοιπόν είναι να υπάρχει μια ενιαία εκλογική περιφέρεια στην οποία ε, θα εκλέγονται οι ευρωβουλευτές. Ο κάθε ε, ψηφοφόρος θα έχει δύο ψήφους. Ε, μία ψήφο για την περιφερειακή εκλογική περιφέρεια και η δεύτερη ψήφος θα αφορά στον ε, ευρωπαϊκό, ε, στην ευρωπαϊκή λίστα υποψηφίων πανευρωπαϊκή. Είναι βέβαια σημαντικό ε, να υπάρχει μια πανευρωπαϊκή εφορευτική, εφορευτική επιτροπή, στην αποκαλέσουμε, που θα ελέγχει την εφαρμογή των, ε, της διαδικασίας και θα καθορίζει τον κανονισμό της διατάξης για την ε, επιλογή και την επικύρωση των υποψηφίων που θα προτείνουν τα πολιτικά κόμματα. Εγώ ε, πιστεύω ότι αυτές οι υπερεθνικές λίστες υποψηφίων ε, θα πρέπει να αποτελούνται από υποψηφίους από διάφορα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να επικρατεί και ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου. Το θέμα τώρα είναι ε, να μεταλλαγούν, να γίνουν τα πολιτικά κόμματα που έχουν τώρα πραγματικά πολιτικά κόμματα. Δεν οργανώνουν απλά συνέδρια όπως κάνουν τώρα, να εντοπίσουν υποψηφίους, να τους βάλουν στις λίστες ε, και να κάνουν ε, εκστρατεία υπέρ των για να εκλεγούν. Αυτό σίγουρα θα οδηγούσε ώστε να είναι πολύ ενδιαφέρον το όλο θέμα για τον τύπο. Θα υπάρχει έτσι η ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος. Και αυτή η διαδικασία ε, θα μπορούσε να εμπλουτιστεί, να γίνει, όλο, να γίνει πιο ενδιαφέρουσα ε, με το να συμπεριληφθούν και επώνυμοι διασημότητες ε, ικανοί διάσημοι άνθρωποι, όχι απλά ηθοποιοί και ποδοσφαιριστές, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ε, προσελκύσει κανείς σε τέτοιου είδους λίστες διασημότητες. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή που προτείνω και αυτό δεν σημαίνει ότι τα εθνικά κόμματα δεν θα μπορούν να ελέγχουν ε, το κοινοβούλιο. Πάντως, ε, πιστεύω ότι αν τελικά επιθυμούμε να έχουμε όρημα ομόσπονδα πολιτικά συστήματα, κάπως έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Και τα πολιτικά κόμματα στις πατρίδες μας ε, θα πρέπει να δεχθούν ότι καλούνται με φιλικό και επικοδομητικό τρόπο να ανταγωνιστούν, γιατί βρίσκονται μέσα σε αυτά τα ομόσπονδα πολιτικά κόμματα, είναι αδελφά κόμματα μιας ευρύτερης οικογένειας. Εν πάση περιπτώσει, τα εθνικά πολιτικά κόμματα που θεωρείται ότι είναι τα οχυρά της εθνικής κυριαρχίας θα πρέπει να αλλάξουν νοτροπία. Εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες επιθυμούν να δουν ότι τα ε, πολιτικά κόμματα προσαρμόζονται. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Βλέπουν ότι δημιουργείται ένταση ανάμεσα ε, στα διάφορα ε, κόμματα σε επίπεδο εθνικό. Και σας το επισημαίνω. Τώρα, Μία πρόταση που αφορά μόνο στα μεγαλύτερα κράτη. που καλούνται ε, στο να έχουν μεγαλύτερες ε, εκλογικές περιφέρειες. Γιατί αυτή τη στιγμή όσο μικρότερη είναι η εκλογική περιφέρεια, τόσο πιο δύσκολο ταυτίζονται οι εκλογείς ε, με τους ε, εκλεγόμενους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ε, να βρούμε κάποια λύση, υποχρώνοντας τα μεγαλύτερα σε έκταση κράτη-μέλη να συστήσουν ε, περιφερειακές εκλογικές περιφέρειες, μεγαλύτερες δηλαδή. Ξέρω ότι αυτό δημιούργησε προβλήματα ε, και πρέπει να συζητηθεί. Σε άλλε χώρε, πρόεδρε, έχουμε ένα κλειστό ψηφοδέλτιο Δηλαδή ουσιαστικά ο ψηφοφόρο εγκρίνει ολόκληρο το ψηφοδέλτιο. Είναι σαν να σταυρώνει όλους τους υποψηφίου. Σε άλλε περιπτώσει πάλι, σε άλλες χώρες, ο ψηφοφόρο μπορεί να επιλέξει υποψήφιο από το ψηφοδέλτιο. Έτσι εκεί μπορεί να ξεχωρίσει ένας ε, πιο δημοφιλής υποψήφιο. στο ισχύ στη Φιλανδία και στο Βέλγιο. Είναι μια προσέγγιση καλή και πιο ελκυστική για τον πολίτη. Να μπορεί δηλαδή να ψηφίσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε διαστολή με την υπερψήφιση ενός απλώς. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα κράτη να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως προείπα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κατανείμουμε τις 751 έδρες του σημερινού κοινοβουλίου μεταξύ των χωρών μας Μπορεί να γίνει αυτό. Επίσης θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε την ψηφοφορία στο Σαββατοκύριακο, γιατί τώρα έχουμε τέσσερις ημέρες στη διάθεσή μας, με αποτέλεσμα που γίνεται στην Ολλανδία, υπάρχει πρόβλημα με την εμπιστευτικότητα. Γιατί στην Ολλανδία δημοσιεύονται τα αποτελέσματα, ανακοινώνται τα αποτελέσματα, Πέμπτη, Παρασκευή, πριν καν ξεκινήσει η ψηφορία στις ε, άλλε χώρε. Και αυτό δεν συνάδει με τις αρχές μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την ε, δραματοποίηση αν η ψηφορία λαμβάνει χώρα. Σε όλες τις χώρες, Σάββατο και ή Κυριακή και μόνο. Μια άλλη πρόταση που έχουμε ξανυποστηρίξει είναι να μετακινηθούν οι εκλογέ λίγο πιο νωρί από τον Ιούνιο, κυρίω για την Σκανδιναβία, και έχουν ένα μικρό καλοκαίρι γύρω από τον Ιούνιο. Οι άνθρωποι θέλουν να απολαύσουν το καλοκαίρι του βεβαίω και, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για να εκλέξουμε κομισιόν τον Ιούλιο, νομίζω ότι η πρόταση αυτή έχει νόημα ειδικά για την Κομισιόν, χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο για να οργανωθούμε εσωτερικά πριν λάβουμε απόφαση την Κομισιόν και τον πρόεδρο της Κομισιόν. Έχουμε επίσης ένα λόγο ζήτημα. Ελάχιστη ηλικία ψηφοφόρων και υποψηφίων. μεγάλης αποκλήσεις και εδώ. Η Αυστριακή. έχουν κατεβάσει το όριο στα 16 έτη. Εγώ το ψηφίζω αυτό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Ο στόχος φυσικά όλες αυτές τις προσπάθειες είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές. Δεν ξέρω αν αυτό το πετυχαίνουμε με την ταπείνωση του ορίου ηλικία, γιατί φαίνεται ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται πολύ για τι εκλογέ, αλλά δεν ξέρω, αξίζει ίσω να το προσπαθήσουμε. Επίση, έχει σε κάθε περίπτωση σημασία να ξαναστείλουμε το μήνυμα στους νέους. Πρέπει επίσης να βοηθήσουμε και να θερύνουμε την πρακτική των υποψηφιωτήτων σε χώρες άλλες από την χώρα προέλευσης του υποψηφίου. σε τόπους οποίους, στον τόπο ενδεχομένω στον οποίο διαμένουν προσωρινά. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει συνεχώ ε, παράπονα από ανθρώπου οι οποίοι είναι στο εντό εισαγωγικών εξωτερικό για κάποιο χρονικό διάστημα και οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία ακριβώ να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογέ. Θέλει έλεγα λοιπόν να ενθαρρύνουμε αυτή τη ε, δυνατότητα και μπορούμε να το κάνουμε. Τέλος. Έχουμε το ακαθόδες ζήτημα των προνομίων και συλλιών των ε, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. το οποίο χρονολογείται από το 1965. Πριν βεβαίως τις άμεσες εκλογές πρώτη για ρύθμιση η οποία δεν ταιριάζει με ένα κοινοβούλιο το οποίο είναι πολύ πιο αυτόνομο σε σχέση με το παρελθόν. Όσοι είναι εδώ μερικά χρόνια γνωρίζουν τις διαμάχες που έχουν ξεσπάσει και στην Ιταλία ή με την Ιταλία. Όσον αφορά το καθεστώς το οποίο διέπει τους ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σχέση και με την εθνική νομοθεσία, η οποία τους καλύπτει. Αυτό δεν θα γίνει εν ε, αυτά ήταν περιληπτικά τα σχολιά μου, οι προτάσεις μου. Και τέλος, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την διαδικασία, θα ήθελα να ολοκληρωθεί η διαδικασία αν δυνατόν τον Σεπτέμβριο, εν συνεχεία να αποστελεί μια στο, στο Συμβούλιο, από το οποίο θα ζητήσουμε να ξεκινήσει τη διακυβερνητική γιατί αυτό απαιτείται για, την, για τις προτάσεις αυτές, πρέπει να τροποποιηθούν οι συνθήκες, έτσι ώστε την άνοιξη του χρόνου να συνεδριάσει η προπαρασκευαστική της διακυβερνητική και βεβαίω τα εθνικά κοινοβούλια, τα πολιτικά κόμματα, η κομισιόν και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να τα συζητήσουν όλα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει και θα είναι δυνατόν να διαμορφώσουμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την διακυβερνητική για να συζητήσουμε μεταξύ άλλων τα θέματα της μεταρρύθμισης αυτής που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να επικεντρωθούμε λοιπόν στις ουσιαστικές ρυθμίσεις της ε, Λισαβόνας. Ε, πιστεύω ότι αυτή η σύνοδος θα μπορούσε να κρατήσει δύο μήνε και θα κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μα του χρόνου το καλοκαίρι. Και εν συνεχεία βεβαίω θα ανοίξει η 12 μήνη περίοδο για την επικύρωση από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έτσι ώστε το 2013 να τεθεί σε ισχύ η σχετική συμφωνία, ώστε να έχουν αρκετό χρόνο τα πολιτικά κόμματα να οργανωθούν εν ώψη των προσεχών, των επομένων ευρωεκλογών του 2014 δηλαδή, με βάση τις νέες ρυθμίσεις. Αυτά ευχαριστώ. Ε, just very... Για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε την έκθεση όπως προτάθηκε από τον Άντριου Ντάφ το Σεπτέμβριο, θα πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις και στις αρχές του Ιουνίου. Η προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών είναι στις 17 Ιουνίου και η ε, ψηφοφορία στην ΑΦΚΟ τον Ιούλιο, λίγο πριν φύγουμε για τις διακοπές μας. Α, να ξεκινήσουμε τον Γεωργιό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νταφ να τον ευχαριστήσω για την έκθεσή του. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι αντιμέτωπο με ένα τέτοιο θέμα. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο αφορά το περιεχόμενο, το δεύτερο αφορά τι διαδικασίε ή μάλλον το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με το πνεύμα αυτής της πρόταση, της μεταρρύθμισης με τη δυνατότητα δηλαδή να προτείνει το Κοινοβούλιο μας, το Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από μια άποψη της αναθεώρησης της, των συνθηκών μία αναθεώρηση του εκλογικού συστήματος. Θα ήθελα να προσθέσω στα όσα ήδη υπόθηκαν και το παρακάτω επιχείρημα. Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο θέλησε είπε ότι η αντιπροσωπευτικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αντιστοιχεί στο μία ψήφος για κάθε άτομο. Αυτό θα μπορούσε να ισχύσει για άλλα εκλογικά συστήματα στον κόσμο, αλλά όχι για το συγκεκριμένο. Σε κάθε περίπτωση βασίζεται σε ένα θέμα αρχής, την δημοκρατική νομιμότητα. Θυμίζοντας αυτή την άποψη του δικαστηρίου της Καλτσρούης, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με αυτό το πνεύμα της ε, πρότασης. Είναι ένα πνεύμα που μας βοηθάει να πάμε πέρα από τα σύνορα, να αποτελέσει, να αποκτήσει η Ευρώπη ένα κόρπους, μια συνοχή. Συμφωνώ λοιπόν με όλα αυτά. Θα πρότεινα ότι ενδεχομένως θα πρέπει να ορίσουμε τη διάσταση της πρότασης. Γιατί εάν θα καταλήξουμε σε μία συμφωνία τη συνθήκης, η συνθήκη, η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να προβλέπει πολλά πράγματα. Αν όμως η πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνει και εθνικές, εκλογικές, βαθιές μεταγνήσεις, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει πιο δυσεπίλητα προβλήματα. Για παράδειγμα, αν ε, αναφερθούμε στην ε, ε, κατώτατη ηλικία των ψηφοφόρων. Τότε θα πρέπει να γίνουν συνταγματικές αλλαγές, κάτι που θα περιέπλεκε ιδιαίτερα τα πράγματα. Θα σας καλούσα λοιπόν να εξετάσετε κατά πόσον η ουσία του θέματος θα έπρεπε να εξεταστεί από την άποψη του εφικτού. Δηλαδή, ένα σημαντικό μέρος των ε, μεταρρυθμίσεων αφορούν μια ευρωπαϊκή λίστα, την έπραξη μιας ευρωπαϊκής λίστας. Ε, και με αυτό συμφωνώ απόλυτα. θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτά που είναι εφικτά και αυτά που δεν είναι εφικτά, γιατί ενδεχομένως δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα. Δεύτερον, θα ήθελα να εκφράσω ορισμένες σκέψεις που αφορούν τη διαδικασία. Μετά ο Ρομπέρτιο Γουαλτέρη που είναι ο σχιώδης εισηγητής της ε, ομάδας μας θα διευκρινίσει το γιατί έχουμε διαφωνίες σχετικά με αυτό το θέμα. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που πρότεινε ο κύριος Νταφ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να προχωρήσουμε με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η μεταρρύθμιση, λαμβάνοντα υπόψη ότι υπάρχει πολιτική δέσμευση μεταξύ των ομάδων, που βασίζεται βεβαίω στη συμφωνία που θα εγκρίνουμε αύριο ή μεθαύριο και που αφορού, αφορά τους νέους 18, 18 ευρωβουλευτές που θα φτάσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και με βάση αυτή τη συμφωνία ξεκινάει αυτή η συζήτηση που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Επειδή όμως θέλουμε να ξεκινήσει μια πρόταση από την Ολομέλεια, αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε μακριά από τις, ε, τα κόμματα, από τις χώρες μας όπου δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτή η συζήτηση είναι κεφαλαιόδου σημασία. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι το να πει κανεί σε μια χώρα σαν την Ισπανία που έχει μια ε, συγκεκριμένη εδαφική πολιτική οργάνωση ότι οι εκλογικές λίστες για τους, ε, τις θα πρέπει να καθοριστούν ε, τοπικά. Αυτό είναι μια απόφαση που δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε εμείς εδώ. Θα προτιμούσα συνεπώς να συνεχίσουμε αφού προηγουμένως συμφωνήσουμε μεταξύ μας, κόμματα, ευρωπαϊκά κόμματα, ε, για να ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται τα όρια. Αυτό θα επιτρέψει στο κοινοβούλιο μας να υποβάλει μια συνενετική πρόταση, μια πρόταση που γίνεται αποδεκτή από το πολιτικό σύστημα. ο τελικός οργανισμός, ο τελικός φορέας θα μπορούσε να δώσει την τελευταία όθηση. Είναι ανώφελο να ετοιμάσουμε ένα έγγραφο και μετά να συγκρουστούμε μπροστά στις πολιτικές, σε μια πολιτική πραγματικότητα που θα εμποδίσει την πορεία αυτής της πρότασης. Θα... Εγώ συμφωνώ απόλυτα με το πνεύμα αυτής της πρότασης. Δίχως άλλο, θα πρέπει να αναλάβουμε δεσμεύσεις για να προχωρήσουμε. Θα έλεγα όμως να επιβραδύνουμε κάπως τους ρυθμούς μας, γιατί έχω πάρα πολλές αμφιβολίες σε ό,τι αφορά πολλές προτάσεις. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι σε ό,τι αφορά τα εκλογικά συστήματα υπάρχουν δέκα χίλιες προτάσεις. Θα, γνωρίζοντας λοιπόν τη σημασία αυτού του θέματος και το διακυβευόμενο καθώς και τα νομικά, συνταγματικά συστήματα που μας περιορίζουν. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα αυτά, θα προτιμούσα να κινηθούμε με βραδύτερους ρυθμούς μεταξύ των άλλων και με βάση μια συνένεση που θα πρέπει να αναζητήσουμε με τις διάφορες χώρες και τα διάφορα κόμματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γουαλτιέρη. Grazie. Ma io devo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 της συμφωνίας ή όχι με την φιλοσοφία και τις προθέσεις του κ. Νταφ, ανεξαρτήτως του αν συμφωνώ ή διαφωνώ, θέλω να πω ότι συμφωνώ. Τουλάχιστον με την φιλοσοφία. Όμως, η πρόταση αυτή δεν μου φαίνεται ρεαλιστική. Διότι προϋποθέτει τροποποίηση των συνθήκων. Και δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένες οι χώρες μας να ξαναδρομολογήσουν μια θεσμική μεταρρύθμιση μετά την επίπονη για και τις οδύνες του το κοιτού της Λισαβόνας. θεωρούμε ότι είμαστε σε περίοδο εφησιασμού και χαλάρωσης και δεν νομίζω ότι χαλάσουν τα κράτη μας τη ζαχαρινιά τους για ένα τέτοιο σκοπό. Γι' αυτό και δύσκολα δούμε αυτές τις προτάσεις του κυρίου Ντάφ να εφαρμόζονται. Είναι μη ρεαλιστικές αυτές οι προτάσεις επιπλέον διότι προϋποθέτουν και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, τροποίηση του ελαχίστου ορίου για το εκλέγεν και το εκλέγεστε. Αυτά πρέπει να γίνουν σε αρκετές χώρες. Και από την ιστορία γνωρίζουμε ότι οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για θέματα εκλογών παίρνουν χρόνια. Με πρώτη τη χώρα μου που συζητούμε παρόμοια θέματα εδώ και 20 χρόνια, χωρίς να έχει επισυμβεί εντωμεταξύ παραμικρή αλλαγή. Εάν κάτι ανθίστε λοιπόν στα συστήματά μας, αυτά είναι τα εκλογικά συστήματα. Πολύ δύσκολα λοιπόν θα καταφέρουμε σε αριθμό χωρών να πετύχουμε τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που αποτελούν και την προϋπόθεση για την υλοποίηση των προτάσεων του κυρίου Νταφ. Ανεξαρτήτως αυτού πάντως, είμαι κάπως επιφυλακτικός ως προς ορισμένες προτάσεις του κυρίου Νταφ. Καταρχήν, η ενιαία ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια, αν και γενικά θα μου άρεσε η ιδέα, φοβούμαι ότι οι περισσότερες χώρες θα την απορρίψουν, διότι θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της εθνικής εκπροσώπησης του σκόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και γνωρίζουμε ότι αυτή θα συνδυαστεί με μια δεύτερη συρρήκνωση λόγω της διεύρυνσης και μόνο, λόγω της εισόδου νέων χωρών. Κάποιοι λοιπόν θα χάσουν έδρες και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Σε πώς πρέπει να επισέλθω στην ουσία των προτάσεων. Επαλαμβάνω ότι έχω τις επιφυλάξεις μου που αφορούν μεταξύ άλλων και την προτιμησιακή ψηφό. Η πρακτική αυτή υπάρχει σε αρκετέ φορέ δεν υπάρχει όμω σε άλλε. Σε αρκετέ. Η προτιμησιακή ψήφο Σταυρό, τουλάχιστον δεν απαιτεί μεταρρυθμίσεις, σημαντικέ τουλάχιστον. Όμως στις χώρες όπου πυλώνε του συστήματος είναι τα κόμματα, η προδημιστική ψήφο, ο σταυρό θα έχει αποτέλεσμα εσωτερικό ανταγωνισμό. Μεταξύ δηλαδή των υποψηφίων του ιδίου κόμματος. Θα είχαμε λοιπόν το φαινόμενο του σφοδρού ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδετών στους κόλπους του ίδιου κόμματος για την εξασφάλιση του σταυρού των ψηφοφόρων. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι η δημοκρατία των κομμάτων. Ψηφίζουμε προτάσεις κομμάτων. Το προσωπικό στοιχείο, πιστεύω, ο Σταυρός θα ανέτρεπε αυτήν την προσέγγιση, αυτήν την φιλοσοφία, το χαρακτήρα των θεσμικών κομμάτων. Αυτό λοιπόν σε εθνικό επίπεδο παραλαμβάνω θα είχε σημαντικέ συνταγματικέ δεν μεταξύ άλλων στη δική μου χώρα και θα ήταν προς πολύ δύσκολο να καλύψουμε σε αποδεκτή ρύθμιση. Τέλος, όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε τις προτάσεις αυτές, παρακαλώ να μην ξεχάσουμε βεβαίω και τον φιλόδοξο στόχο, αλλά και τους εγγενείς περιορισμούς και την σύνεση που απαιτείται για τους σκοπούς αυτής της συζήτησης. Κύριε Νταφ, μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε τα πάντα αν θέλετε. Όμως να μην ξεχάσουμε ότι τα περιθώρια που έχουμε, τα τέσσερα προσεχή έτη, να ε, μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα οποία είπε ο κύριος Νταφ, τα περιθώρια αυτά είναι πολύ στενά. Δεν ε, θέλω να εκλειφθεί στάσιμος υπερβολικά ε, διστακτική. Χρειάζεται όμω σύνεση σε κάθε περίπτωση. Θεωρώ απλώ ότι οι πολιτικέ προποθέσει δεν συντρέχουν να μπορέσουμε να πετύχουμε τον φιλοδόξο πολιτικό στόχο του κ. Νταφ εντό τη παρουσία εντολή. Κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα προσθέσω πολλά στα όσα ήδη υπόθηκαν. Και για τον λόγο αυτό η παρέμβασή μου θα είναι σύντομη. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Νταφ στην αρχή της παρουσίασής του. Εξέφρασε κάποια αμφιβολία. Είπε ποιος ξέρει αν ενδιαφέρει το θέμα αυτό τους βουλευτές. Βασίστηκε στο γεγονός ότι πολύ λίγοι από μας είναι παρόντες από τις παρεμβάσεις όμως που έγιναν, ο κύριος Ντάφτα πίστηκε ότι το θέμα αυτό ενδιαφέρει πολλούς από εμά. Κατάλαβα τι εννοεί ο κύριος Ντάφτ και θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τα επιχειρήματά του, συμφωνώ με το όραμά του. Θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα όριμα που εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη από το Ηνωμένο Βασίλειο προέρχεται μία τόσο φιλοευρωπαϊκή άποψη που αφορά την πολιτική εκπροσώπηση, τις διαδικασίες για να υπάρξει αυτή η πολιτική εκπροσώπηση. Θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ και με μερικές από τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν γιατί πιστεύω μεταξύ των άλλων ότι υπάρχει κάποια κόπωση σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη. Η πορεία που ακολουθείται είναι μακρά, είναι κουραστική, αλλά παράλληλα Είναι αλήθεια ότι η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στα εκλογικά συστήματα των μεμονωμένων χωρών είναι κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Υπάρχουν πολλές κόρες στις οποίες γίνεται αναφορά στις εκλογικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών. Θα ήθελα να πω όμως ότι μπήκε μια τροχοπέδη σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το πλειοψηφικό στον ολογικό, ε, η εφαρμογή του συστήματος της προσημητιακής ψήφου σε άλλες χώρες μιλάνε για άλλες μεταρρυθμίσεις. Αν λοιπόν υπήρχε η δυνατότητα εφαρμογής του, μιας μεταρρύθμισης του εκλογικού συστήματος για τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι μεταρρυθμίσεις αυτές τα συνέβαλαν στο να έρθουν στην επιφάνεια προβλήματα και να δημιουργηθεί μία αντίσταση σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι ανοίγουν την πόρτα και για άλλες μη συνενετικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις εκλογές. Εμείς δεν είναι ότι δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να εντοπίσουμε το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες για να προσθέσουμε, ε, να προσθέσουμε μια συμφωνία που να αφορά τις ημέρες διεξαγωγής των εκλογών. Και αυτό είναι ένα ε, μείζον θέμα. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ευρώπη Ευρωπαίοι πολίτε ψηφίζουν για τι ευρωεκλογέ την ίδια μέρα είναι κάτι που στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Επίση, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά την ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων. Ορισμένε χώρε το προβλέπουν στην ομοθεσία του, άλλε χώρε πάλι όχι. Και πιστεύω ότι θα ήταν δυνατό να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για να γίνουν το Μάιο οι εκλογέ για του λόγου που παρέθεσε ο κύριο Ντάφα για λόγους που αφορούν τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Σε ό,τι αφορά τα προαπαιτούμενα επίσης θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία, αλλά και για τα εκλογικά κατόφια θα μπορούσε να βρεθεί μια συμφωνία. Πιστεύω ότι θα, μπορούσε, ε, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και για ένα ποσοστό ευρωπαϊκά, από ευρωπαϊκές λίστες και όχι εθνικές λίστες. Τώρα, για το θέμα της ηλικίας των ψηφοφόρων, της κατώτητης ηλικίας των ψηφοφόρων. Ενδεχομένω θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια συμφωνία. Θα μπορούσαμε να καταβάλουμε μια προσπάθεια. Πιστεύω όμω ότι θα είναι πολύ δύσκολο και οι 27 χώρε να δεχτούν ένα ενιαίο σύστημα κοινών εκλογικών περιφερειών ή ένα ε, κοινό σύστημα υπολογισμού των ψήφων. Δεν θέλω να πω ότι αυτός είναι ο επιθυμητός στόχος Ενδεχομένως 21 θα μπορούσαν να συμφωνήσουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχουν εθνικές εκλογικές περιφέρειες. Αυτό όμως θα μπορούσε να εφαρμοστεί αν συμφωνήσουν 27 28 χώρες μέλη αν υπολογίσουμε και την Κροατία. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει στόχος μας να είναι ή όλα ή τίποτα θα πρέπει να εντοπίσουμε τα στοιχεία εκείνα που κατά την άποψή μας θα μπορούσαν να είναι εφικτά, να δώσουμε τη μάχη μας, να δώσουμε τη μάχη μας ακόμα και για το ανέφικτο. Θα μπορούσε όμως να υπάρξει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Καλύτερα να κάνουμε πέντε, τέσσερα, τρία μικρά βήματα, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση, αντί να κάνουμε, να δώσουμε ε, ένα πίδο στο απόλυτο σκοτάδι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στρασκόφσκι, ο αντιπρόεδρος. Α, δικηγόρος... Ως δικηγόρος ε, του Λαδιαβόλου θα μιλήσω για τις 25 ε, χώρες μέλη των ψηφίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξετάζοντας τα διάφορα συστήματα στις διάφορες χώρες, το πρόβλημα είναι ότι αν δεν υπάρχει μία λίστα κλειστή, κλειδωμένη σε μία συγκεκριμένη χώρα, οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι είναι απόμακροι οι άνθρωποι αυτοί και δεν έχουν καμία σχέση με την εκλογική τους περιφέρεια. Έχουμε τα προβλήματα αυτά ακόμα και σε περιφερειακές εκλογές, με ανοιχτές λίστες. Τα συστήματα αυτά είναι από μία άποψη καλύτερα, γιατί είμαστε πιο κοντά στην εκλογική μας περιφέρεια. Νομίζω ότι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι να εκλεγεί κάποιος και να εξαφανιστεί στις Βρυξέλλες και να μην το ξαναδεί κανένα η εκλογική του περιφέρεια τα επόμενα πέντε χρόνια. Και πάλι μιλάω ως δικηγόρος του διαβόλου. Καταλαβαίνω το λόγο ύπαρξης αυτής της λίστας, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να εκλέγουμε άτομα από αυτές τις λίστες και να μην τους ξαναδούμε ποτέ πια στις χώρες μας. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει αυτή την αίσθηση της αποξένωσης. Καταλαβαίνω τι λέτε με όλες αυτές τις διασημότητες που τους εκλέγουμε και μετά δεν τους ξαναβλέπουμε. Θα μπορούσε το αποτέλεσμα να είναι αντιπαραγωγικό. Οι άνθρωποι θα περιμένουν κάτι να συμβεί και μετά θα απογοητευτούν. Έχω συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν την ιδέα σας. Καταρχάς, όταν περάσουμε στη φάση των εκλογ, της εκλογής αυτών των ανθρώπων με βάση αυτές τις λίστες, ε, τι, πού θα βασιστούμε, θα γίνει μια στάθμιση, θα γίνει καταμέτρηση των ψήφων, θα λάβουμε υπόψη πρωτοβουλίες των πολιτών. Πώς θα γίνει, θα εκλεγεί αυτός που έχει η το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων ή θα συνυπολογιστεί το, η χώρα από την οποία προέρχεται. Θα υπάρξει ένα επιπρόσθετο στοιχείο που θα περιπλέξει τα πράγματα. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένε Πολιτείε δεν ξέρει καλύτερα ε, ε, τα περί εκλεκτόρων. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό το πώς κάποιος που παίρνει μικρότερο αριθμό ε, ψήφων εκλέγεται. Γιατί αυτό που μετράει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ψήφος των ελεκτόρων. Αυτό θα μπορούσε όμως να παραπλανήσει ανθρώπους που θα δεκτούν αυτή την ιδέα. Το δεύτερο ερώτημα. Προβλέπετε κάποιος που βρίσκεται σε μία διακρατική λίστα να είναι και σε μια εθνική λίστα. Θα μπορεί κανείς παράλληλα να συμμετέχει σε δύο λίστες. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ε, προβληματικό, ας πούμε, όταν μιλάμε ε, για αυτούς τους διάσημους που είπατε και οι οποίοι θέλουν να έχουν εγγύησει ότι θα εκλεγούν. Απ' την άλλη πλευρά, το να είναι κανείς σε δύο λίστες δεν ξέρω είναι καλή ιδέα. Οι κατάλογοι αυτοί, οι λίστες αυτές θα πρέπει να είναι ανοιχτέ, να είναι κλειστέ για να υπάρχει πραγματική επιλογή υποψηφίων. Ύστερα υπάρχει το θέμα της χρηματοδότησης. Θεωρώ ότι η εκστρατεία για αυτές τις διακρατικές λίστες θα οργανωθεί από τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά κόμματα θα πληρώσουν το κόστος αυτών των εκστρατιών. Εγώ απλά και μόνο εστιάζω την προσοχή μου σε αυτά τα προβλήματα για να μπορέσετε να το σκεφτείτε. Το θέμα της χρηματοδότησης. Όπως ξέρετε τώρα δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις εκστρατείες μας από ευρωπαϊκά κονδύλια εκ το Μάρτιο και μετά είναι δικό μας θέμα. Αν θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε αυτή την αίσθηση, την πανευρωπαϊκή, τότε αυτές οι εκστρατείε θα πρέπει να κινηθούν εκ παραλίλου. Δηλαδή, ο συμμετέχων στην διακρατική λίστα έρχεται στη Βασοβία, στη Μαντρίτη, κάνει την εκστρατεία του και παρουσιάζει τους υποψήφιους από την εθνική λίστα για να μπορέσουν να συγκεραστούν όλα αυτά. Δηλαδή ε, ο διακρατικός υποψήφιος να συνεργάζεται κάτω, μέσα στο ίδιο πλαίσιο με τους εθνικούς υποψήφιους. Είναι όμως εδώ ε, θέμα χρηματοδότησης, γιατί θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου θα ε, δώσει κανείς ιδιαίτερη βαρύτητα σε ορισμένους τομείς. Δηλαδή, σε μία πρώτη φάση να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε για τα προβλεπόμενα, για τα επερχόμενα και να, μετά να μην μείνουν χρήματα για άλλα. Τώρα, εάν υπάρχει αυτή ε, η, η, η τότε θα είναι άδικο για ορισμένους. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά τα θέματα. Okay, thank you very much. If uh, you allow me, then I also would like to make some comments. So first of all, uh, you, you, you, you... Κοιτάξτε, Πρώτα απ' όλα, από το 99 ξέρετε ότι είναι ο κύριος Αντάφα στο Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου, επειδή είναι αρκετό καιρό εδώ σε αυτήν την Επιτροπή, επιθυμεί να θεσπιστεί νομοθεσία που θα είναι καλή για τους ε, Ευρωπαίους ε, πολίτες. Και είμαι σίγουρη ότι ε, θα αναπτύξετε πολλές επαφές και έχετε επαφές όχι μόνο με τους ε, πολιτικούς ε, ομοειδεάτες σας, αλλά και με τις ΜΚΟ. Το τουλάχιστον έγινε κατά το παρελθόν. Ε, στην έκθεσή σας αναφέρετε ότι από το 63% το 70 τόσο έπεσε στο 43% τις τελευταίες εκλογές. Αυτό αφορά την συμμετοχή στις εκλογές και πράγματι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγεται. Εγώ πιστεύω ότι η άποψή σας να υπάρχουν ευρωπαϊκά κόμματα και να υπάρχουν και ευρωπαϊκά ιδρύματα, σε αυτό το σκεπτικό καταλήγουμε ότι χρειαζόμαστε και ευρωπαϊκούς αριθμούς συνάδελφοί μου έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις ε, και νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή που ξεκινήσαμε. Πιστεύω λοιπόν ότι οι επιπρόσθετοι 25 ευρωβουλευτές θα έδραν και άλλη, άλλη εικόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε 35% γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς ε, το θίγετε το θέμα αυτό στην έκθεσή σας. 24% είναι ο μέσο όρο ε, γυναικών, ποστό γυναικών ε, στα εθνικά κοινοβούλια. Σε κάποια όμως κοινοβούλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε κάτω από 10% γυναίκες στο σύνολο των βουλευτών. Γι' αυτό θεωρώ ότι επειδή είμαστε το 52% ε, του πληθυσμού ε, πρέπει να έχουμε καλύτερη εκπροσώπηση και το θεωρώ ότι εγώ είμαι πολύ τυχερή που είμαι εδώ αντιπρόεδρος σε αυτήν την επιτροπή ως γυναίκα. Εσείς βέβαια κύριε Ραφάλ είστε ο μόνος που εξέφρασε την άποψη ενός μεγάλου ευρωπαϊκού οικονόματος. Γι' αυτό λοιπόν ε, πιστεύω ε, τι πιστεύουν ε, και οι ε, συναδελφοί σας στο ίδιο κόμμα. θα καταλαβαίνετε βέβαια ότι εγώ προσπαθώ να είμαι δίκαιη και θέλω να μιλήσουμε για την έκθεση και για τα συμπεράσματά της. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε αυτό το θαυμάσιο σχέδιο. Αυτά είναι τα δικά μου τα σχόλια και θα ήθελα να ρωτήσω ότι ε, σας προκάλεσα λιγάκι, αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψη και μιας ε, άλλης γυναίκας και μετά θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Νταφ για να κάνει ε, τα τελικά του συμπεράσματα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Νταφ. Ο λόγος τον οποίο δεν ζήτησε τον λόγο είναι η καθυστέρησή μου, για λόγους ανεξαρτήτως της θέλησή μου, για μια συζήτηση πολύ σημαντική κατά τα άλλα. Συγγνώμη λοιπόν που δεν ήμουν εδώ και δεν μπόρεσα να παρουσιάσω το απόψη μου νωρίτερα πάνω στην εργασία του κύριου Νταφ. Το θέμα μας είναι πολύ σημαντικό. Η εμπέδωση της δημοκρατίας και η αντιπροσωπευτικότητα στην Ευρώπη. Δεν έχω μεγάλη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως άλλα μέλη απέδειξαν με τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους στην ε, Επιτροπή αυτή. στους κόλπους του ΕΛΚ, ε, άλλωστε ούτε εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αν το βάθη. Αυτές τις ε, ιδέες ε, του κυρίου Νταφ που χαρακτηρίζονται από εφαιρετικότητα και καινοτομία. Θέλω λοιπόν να πω, απαντώντας στον κύριο Νταφ και στους συναδέλφους, ότι πρέπει να εμβαθύνουμε στο θέμα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε άπρακτοι στην συρρυκνωμένη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωεκλογέ. Άλλωστε αυτό άπτεται της δημοκρατικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να παραμένουμε άπρακτοι, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε λύσεις. Συμμερίζουμε επίσης τον ε, ρεαλισμό ορισμένων από τους πολλαλήσαντες. μπορούμε να ξεχνούμε ότι μόλις έκλεισε μια επίπονη φάση θεσμικής αναθεώρησης που δυσκόλυψε ορισμένες χώρες. ασχόλησε τους πολιτικούς, τα πολιτικά κόμματα, τους ε, πολιτισμούς, μας, όσους ενδιαφέρονται, εν πάση περιπτώσει, από την εξέλιξη των ευρωπαϊκών θεσμών. Το κεφάλαιο αυτό κράτησε σχεδόν 10 χρόνια, μόλις έκλεισε. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν συνετό να ζήσουμε για λίγο τουλάχιστον την εφαρμογή της συνδίκης της Λισαβόνας να χωνέψουμε αν θέλετε τις τελευταίες εξελίξεις πριν δρομολογήσουμε ένα νέο θεσμικό κεφάλαιο το οποίο πιθανώ θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσει. Πραγματικά, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσαν η ε, κοινή γνώμη στη χώρα μου, για παράδειγμα, εάν άκουγαν για άλλη μία θεσμική μεταρρύθμιση, τα οποία δεν ξέρω πώς θα καταλάβουν, όπως άλλωστε δεν κατάλαβαν και πολλά από την προηγούμενη. Λοιπόν, έκκληση σε σύνεση και ρεαλισμό. δεδομένων και των δυσκολιών να κλείσουμε το προηγούμενο θεσμικό κεφάλαιο. Ούτως ή άλλως η νέα συνθήκη για αλλαγές όσον αφορά τα προνόμια και τις μας. Ας τα δούμε λοιπόν πώς εφαρμόζονται στην πράξη. Δεν ζούμε σε ένα ιδανικό κόσμο, αυτό είναι βέβαιο. Ας τα ζήσουμε λοιπόν λίγο στην πράξη και ας δούμε σιγά σιγά τι βελτιώσει μπορούμε να επιφέρουμε και πώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν μπορούμε να βελτιώσουμε συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένε πτυχέ όλων αυτών, ε, χωρί να αλλάξουμε τα πάντα εκβάθρων. Α κάνουμε λοιπόν θετικά βήματα, συγκεκριμένα μικρά βήματα προ τα εμπρό, επικοδομητικά. Να εξασφαλίσουμε σίγουρα καλύτερη αντιπροσώπευση των γυναικών, γιατί όντω δεν υπάρχει υποχρέωση ίσης εκπροσώπησης στις εκλογές. Αυτό ε, πρέπει το, το μήνυμα να το στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε εννοείται για την εντονότερη εκπροσώπηση των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να συμπαρθούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, μια άλλη καλή ιδέα που συζητούμε εδώ και καιρό είναι ναι, να συγκεντρωθούν οι εκλογές τις ίδιες μέρες. Οι εκλογές να γίνονται την ίδια μέρα, αν γίνεται, ε, κάτι το οποίο εξευρωπαίζει λίγο περισσότερο, αν θέλετε, τις εκλογές. Αυτά είναι κάποια μικρά πρακτικά πράγματα τα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα μπορούμε να τα περάσουμε σε όλες τις χώρες. Και αυτό σίγουρα θα έστελνε ένα πιο ευρωπαϊκό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε σύγκριση με σκέψεις ε, που αφορούν το απότερο μέλλον όσον αφορά την νομιμοποίηση δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα χρειαστεί λίγο περισσότερο, χρόνο, χρόνος για αυτά νομίζω από την κοινή γνώμη στις χώρες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το, θα πρέπει να είναι το Μάιο. Βεβαίως. Είναι καλή αυτή η ιδέα. Σας ευχαριστώ πολύ, ιδιαίτερα για όσα είπατε για τις γυναίκες. Ο κύριος Ντάφη. Στις CBC στο 322 θα γιορτάσουμε την 60η επέτειο από την διακήρυξη του Σουμάν και καλούνται, καλείστε όλοι να παρακολουθήσετε. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα αν θα μπορούσατε να έρθετε και να μπορέσει να γίνει μια συζήτηση για τα σημαντικά αυτά θέματα. Θα ακολουθήσει ποτό, κάτι που είχε πάντοτε αρκετά ελκυστικό. Θα πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει η τέλεια εκλογική διαδικασία. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Εδώ δεν αναζητάμε την τελειότητα ή την καθαρότητα. Το μόνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε μία κατάσταση η οποία σαφώς απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική. Αυτό είναι κάτι που δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε τα προηγούμενα 12 χρόνια. Θα μπορούσε κανείς να ακολουθήσει τα όσα είπαν μερικοί συνάδελφοι ε, και να πιστέψει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να το αποφασίσει αυτό το θέμα. Είναι δύσκολο να βρει κανείς μια ισορροπία μεταξύ του να αναζητάει, να επιβάλλει ένα κοινό σύστημα και το να αναζητάει το σεβασμό του κοινών αρχών. Και στην πρόσταση μου προσπαθώ να κάνω και τα δύο. να συμβάλλω έτσι ώστε τα συστήματα, τα ισχύοντα συστήματα να ε, ε, είναι περισσότερο κοντά στις κοινέ αρχές και να επιβάλλω την ιδέα μιας διακρατικής εκλογικής περιφέρειας η οποία θα οργανωθεί και θα αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από αυτό το επίπεδο. Από το επίπεδο το δικό μας. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να τρομάξει μερικούς. Εγώ θα τους ενθάρρυνα να δείξουν λύτερη τόλμη. Και ο χώρος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι στα πλαίσια μιας σύμβαση. Θα πρέπει να πω ότι υπάρχει, είναι ένας ε, χώρος έκφρασης ε, πολλών ιδεών, ανταλλαγής πολλών απόψεων, είναι μια πραγματική πρόκληση σε επίπεδο διανοητικό, πνευματικό. Είναι ένα πολύ γόνιμο έδαφος και εκεί συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Όσοι δηλαδή ενδιαφέρονται για τη μεταρρύθμιση αυτής της κλίμακας που προτείνω. Όλοι θα συμμετέχουν σε μια τέτοια άσκηση. Δεν θα πρέπει κανείς να φοβάται ότι κινούμεθα με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Γιατί αυτό που κάνουμε από την απαρχή κιόλας αυτής της πρότασης είναι να αναφερθούμε στη διακυβερνητική σε τελευταία ανάλυση η διακυβερνητική αποφασίζει και οι χώρες θα πρέπει να συμφωνήσουν. Οι Ισπανοί δηλαδή που φοβούνται για τις αυτόνομες εκλογικές περιφέρειες θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τους φόβους τους. Και η διακυβερνητική Γι' αυτό υπάρχει. Αν στο τέλος των συζητήσεων η Ισπανία δεν έχει ικανοποιηθεί με την πρόταση, θα μπορούσε να αρνηθεί, να μην εγκρίνει ένα κομμάτι από αυτή την πρόταση. Αυτή είναι η, διαδικασία που προτείνω και συνιστώ. Δεν θα πρέπει λοιπόν να, να θεωρήσουμε ότι εξωθούμεθα το να πάρουμε αποφάσεις που μετά θα μετανιώσουμε. Υπάρχει αρκετός χρόνος για εκτενείς διαβουλεύσεις που να αφορούν το ίδιο της κοινοβουλευτική δημοκρατίας που θέλουμε. Ένα-δυο σημεία ακόμα. Η Καλιστρούη αναφέρθηκα στην επεξηγηματική, ζευγικό σημείωμα στην απόφαση του δικαστηρίου. Είχα ήδη μιλήσει για αυτό το θέμα, ήταν μια πολύ κακή απόφαση. Παρόλα αυτά, το λογικό, το, η λογική, το σκεπτικό της απόφασης είναι αρκετά ενδιαφέρον και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κριτική που έχει γίνει σε ό,τι αφορά την παρούσα σύνθεση του Κοινοβουλίου καθώς και την άποψη του Γερμανικού Κοινοβουλίου ότι η Γερμανία πλήττεται από την αρχή, αφήγεται από την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι απόλυτα κατανοητό. Εγώ συμπληρώνω τις εθνικές αντιπροσωπείες με 25 συμπληρωματικούς βουλευτές. Δηλαδή, εμείς δεν προσπαθούμε να περικόψουμε από την ποσόσωση της κάθε χώρας. Δίνουμε αντίθετα στους πολίτες την δυνατότητα να έχουν μια εκτεταμένη πρόσβαση, μια μεγαλύτερη ευθύνη να προωθήσουν τις πολιτικές τους επιλογές μέσα από την εκλογική αυτή περιφέρεια των 27 κρατών. Είναι πιθανό σε μεταξύ αυτών των βουλευτών να είναι και Γερμανοί. Αυτό το λέω στην ετότητα. Είναι πιθανόν. Μερικές, μεταξύ αυτών των επιπλέον 25 βουλευτών μπορεί να υπάρχουν και Γερμανοί. ως ένα βαθμό αυτή είναι μία απάντηση στο πρόβλημα που έθεσε το δικαστήριο της Καλσρούης. Ωραία, έθιξε μερικά συγκεκριμένα θέματα. Όχι, δεν προβλέπω ότι η ψηφοφορία για τις διακρατικές ε, λίστες καθοριστεί από την κάθε χώρα, δηλαδή μία ψήφος για κάθε πολίτη. Η διακριτική ευχέρεια έχει με το ότι δεν είναι υποχρεωτικό να δεχτείτε ένα δεύτερο ψηφοδέλτιο πριν περάσετε στην κάλπη. Αν ψηφίσετε, όμως, Μία εστονική ψήφος θα μετράει το ίδιο με μία γαλλική ψήφο. Είναι δυνατόν για ένα βουλευτή, για ένα υποψήφιο να βρίσκεται σε δύο λίστες. Αυτό είναι ένα θέμα που θίγω στο επεξηγηματικό μου μνημόνιο. Η πρακτική διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη. Σε ορισμένες χώρες μπορεί κανείς να είναι υποψήφιος σε δύο εκλογικέ περιφέρειες ε, κατά τον ίδιο χρόνο. Και εάν εκλεγείτε μπορείτε να επιλέξετε ποια θα εκπροσωπήσετε, την εκλογική περιφέρεια Α ή Β. Σε άλλες χώρες η σκέψη και μόνο ότι μπορεί κανείς να βρίσκεται σε δύο μέρη κατά τον ίδιο χρόνο είναι ένα ανάθεμα. Θα πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα. Θα πρέπει να δούμε εάν μπορούμε να επιτύχουμε μία συνένεση που θα ικανοποιήσει όλους μας. Μπορεί να μπορούμε, μπορεί και να μην μπορούμε. Το θέμα της χρηματοδότησης. Βεβαίως είναι απαραίτητο να αλλάξει ο κανονισμός για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Κατά την άποψή μου είναι παράλογο είναι ανόητο το να θελήσουμε να εμποδίσουμε τα πολιτικά κόμματα από το να οργανώνουν τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Τώρα ε, το που γίνεται είναι να υπάρχουν πανό, να κινούνται μέσω ίντερνετ. Αυτό μπορούν να κάνουν. Εγώ προσπαθώ να τα αλλάξω τα πράγματα. να επανέλθουμε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Να υπάρξει μια διασύνδεση μεταξύ των πολιτών και των αρχών εδώ στις Βρυξέλλες που ασκούν την εξουσία. Να μπορούν εδώ οι βουλευτές να εκφράζουν τις, τα όνειρα των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Αυτό χρειαζόμαστε, αυτό δεν υπάρχει. Και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε ελκυστικά και ισχυρά κόμματα είναι μόνο με διακρατικές λίστες. Όλη η ιδέα ότι η Ομοσπονδία του ΕΡΤ θα γίνει κάτι καλύτερο κτλ. Αυτά είναι ανοησίες. Τα δοκιμάσαμε αυτά. Όλα τα κόμματα τα δοκίμασαν. Δεν λειτουργούν όμως αυτά. Δεν οδηγούν σε ανάπτυξη. Δεν καταφέρουν να σταθούν στο ύψος των δημοκρατικών προκλήσεων με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωπες και, αντιμέτωπες και που αφορούν την νομιμότητα. Και αυτό είναι ένα θέμα που προσπαθώ να επιλύσω. Είμαι ευγνώμων σε όσους μίλησαν, αρκεί αρκετοί σοσιαλιστές από τον Νότο. Δεν έχω τίποτα κατά του Νότου ή των σοσιαλιστών. Θα πρέπει να συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή την ευκαιρία να διευρύνουμε την βάση μας. Αυτό ας το συμπεριλάβουμε την ημερησία διάταξη της επόμενης συνάντησης, πρώτο θέμα στην ημερησία διάταξη, έτσι ώστε να είναι όλοι παρόντες και να ασκήσουν τα καθήκοντα που έχουν ως υπεύθυνα μέλη αυτής της Επιτροπής. Δεν είναι απαραίτητο να είναι το πρώτο θέμα στη μερίσια διάταξη. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε όλους εσάς ε, που κάνατε τα σχόλια για αυτό το σχέδιο της έκθεσης και από ό,τι ξέρετε και ξέρω, ε, τέλειωσε ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε τη δουλειά σας, ευχαριστούμε τους ε, διερμηνείς και σας εύχομαι καλό μεσημεριανό διάλειμμα με γεύμα και καλό απόγευμα. Γεια σας.